Πρέπει να σας πω επίσης ότι θα ακολουθήσουμε διαφορετική σειρά στην ημερήσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Μακάρθη, εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξη ραγώγηση στη συνέχεια ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την προληπτική εποπτεία πιστοτικών ιδρυμάτων. Μπορούμε να εγκρίνουμε τις αλλαγές αυτές στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ανακοινώσει της Προέδρου μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης, κανονισμός και οδηγία όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την Ερλίν Μακάρθη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε προκειμένου να περάσουμε σε κάποιες από τις λεπτομέρειες εργασίας που έχω επιτελέσει. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα σχόλια τα οποία έκανα αρχικά. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τα ζητήματα της κατάχρησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει πλέον έναν κανονισμό περνώντας από την απλή οδηγία που είχαμε το 2003 και έχουμε όμως και μία επιπλέον οδηγία όσον αφορά τις ε, κυρώσεις που μπορούν να προβλέπονται. Είμαστε υπέρ λοιπόν της αναβάθμισης της ενίσχυσης ε, του πλαισίου για την καταπολέμηση της κατάχρησης της αγοράς. Στο διαθέσιμο χρόνο που έχουμε θα ήθελα να σας προτείνω κάποιες από τις αλλαγές που έχουν γίνει στην έκθεσή μου. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν εμένω στα σημεία αυτά τα οποία έχω εισάγει στην έκθεση αυτή. Απλώς σας λέω ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να διασαφινιστούν, κάποια σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Έχω συζητήσει και με τους κοιόδης εισηγητές και προσβλέπω σε μια έγκριση του κειμένου που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Θα ήθελα να αφαιρθούμε σε κάποια από τα ζητήματα αυτά και χαίρομαι που είναι και ο κύριος Φέμπερ εδώ παρόν, γιατί είναι εισηγητής για το ΜΥΦΗ, την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός με την δική του οδηγία, με το πλαίσιο το οποίο αυτός έχει αναλύσει την έκθεσή του γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Μία από τις βασικές αλλαγές που έχω κάνει στην τροπολογία παριθμών 1 είναι ότι δεν έχουμε πλέον την κατηγορία OTF, δηλαδή για, τις οργαν... για τους οργανωσμένους μηχανισμούς διαπραγματεύσεων. Δεν γνωρίζαμε ακριβώ τι θα κάναμε με την κατηγορία αυτή πρωτού υποβληθεί η οδηγία MIFID. Ωστόσο, με τις συζητήσεις που είχαμε τους ρυθμιστές, με τις ρυθμιστικές αρχές, ουσιαστικά κατέδειξαν ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός της αγοράς, ότι υπάρχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά διαφορετικά μέσα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, πράγμα το οποίο οδηγεί με τη σειρά του σε όλο και περισσότερα φαινόμενα κατάχρησης της αγοράς. Όταν πήγαμε στη Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κονγκ πρόσφατα, ήταν ξεκάθαρο ότι οι ασιατικέ αγορέ δεν είναι τόσο κατακρεματισμένε οι ευρωπαϊκέ αγορέ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η εποπτεία στην περιοχή αυτή είναι λιγότερο πολύπλοκη και καταφέρουν να καταπολεμήσουν καλύτερα τα φαινόμενα κατάχρησης αγοράς. Η τελική απόφαση για το αν θα πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία για το σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί στα πλαίσια της έκθεσης Φέρμπερ. Εγώ πάντως στην έκθεσή μου τονίζω ότι η δημιουργία όλων και περισσότερων μέσων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερο κατακαιρματισμό που με τη σειρά του οδηγεί σε μεγαλύτερα φαινόμενα κατάχρησης της αγοράς. Είναι σαφές πάντως ότι ε, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε σε μια ξεχωριστή κατηγορία για πλατφόρμες διαπραγμάτευσης. Τώρα, όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες, τις σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες. Έχω χρησιμοποιήσει κάποια εκτιμώντας από προηγούμενες ε, οδηγίες για την κατάχρηση της αγοράς, όπου θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια σημεία για να ορίσουμε με καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο νοούμε λέγοντας insider dealing και εμπιστευτικές πληροφορίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα μία νομική ασφάλεια υπήρχε ένα νομικό ζήτημα με μια, έναν ευρύτερο ορισμό των εσωτερικών επιστευτικών πληροφοριών που πάλι τα ενδιαφερόμενα μέρη εδώ πέρα μας είπαν ότι δεν υπήρχε κάποια νομική σαφήνεια ως προς το αν κάποιες πληροφορίες ήταν σημαντικές ή όχι ή αν για παράδειγμα κάποιες συνομιλίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Φοβόντουσαν με άλλα λόγια ότι μπορεί να εγκριθούν πάρα πολύ αυστηροί κανόνες που να μην επιτρέπουν καμία ανταλλαγή ή χρήση πληροφοριών. Όπω είπα και σε προηγούμενη συζήτηση που είχε γίνει, δεν θα διαγράψω το σημείο αυτό από το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μολονότι καταλαβαίνω το Συμβούλιο οδεύει ουσιαστικά προ μία διαγραφή. Πιστεύω πάντω ότι ε, δεδομένων των συζητήσεων που είχαμε με τους ρυθμιστές, η ε, κατάχρηση αγοράς είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Χρειάζεται ένας ευρύτερος λοιπόν ορισμός για τους ρυθμιστές Χρησιμοποιώ λοιπόν εδώ πέρα μια διατύπωση που πιστεύω ότι αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης και να οδηγήσουν σε κατάχρηση της αγοράς. Άρθρο 6 παράγραφος ε Συζήτησα με το σημείο αυτό κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Ουσιαστικά στο σημείο αυτό προσπαθώ να αποσαφηνίσω με έναν καλύτερο τρόπο τι πληροφορίε αυτέ, καθώ επίση και την χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών αυτών και πώς μπορούμε βάσει της χρήσης αυτής να κρίνουμε αν η συμπεριφορά του φορέα που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές είναι σωστή ή όχι, αν μπορεί να αποτελέσει δηλαδή περίπτωση κατάχρησης αγοράς ή όχι. Όσον αφορά τώρα την εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Κάθε φορά έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να επιβαρύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ένα ιδιαίτερα υψηλό άχθο γραφειοκρατικό. Αυτή τη στιγμή όμω δεν μιλάμε για γραφειοκρατικό άχθο, δεν μιλάμε για διοικητικό άχθο, μιλάμε για κατάχρηση τη αγορά και για την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Έγινε μία απόπειρα να δημιουργηθούν κάποιες εξαιρήσεις ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις ίδιες ακριβώς απαιτήσει. Εγώ διέγραψα πάντως τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει παρέκκληση για τις επιχειρήσεις αυτές και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Βιοτεχνιών λένε ότι και οι ίδιες θεωρούν ότι χρειάζεται να υφίστανται οι ίδιοι κανόνες και για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουν ουσιαστικά να εξαιρεθούν από τον κατάλογο που προβλέπετε. Δεν ξέρω τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρόκειται να κάνει, θα προχωρήσει σε εξαίρεση ή όχι. Αν δούμε τώρα τις υφιστάμενες ε, τάσεις που υπάρχουν σε διάφορες ε, επιχειρήσεις ε, επενδύσεων και παροχής συμβουλών, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι brokers που λειτουργούν όλο και περισσότερο à carte. Μπορεί να έχουν, ε, για παράδειγμα, κάποιες πολύ μικρές, μπορούν να έχουμε κάποιες πολύ μικρές επιχειρήσεις με 10 για παράδειγμα μόνο εργαζομένους που μπορούν να διαχειρίζονται όμως τεράστια ποσά. Η JP Morgan παρουσιάζεται ως μια μικρή επιχείρηση αυτή τη στιγμή Μπορεί να έχουμε και τραπεζίτες ή επενδυτές οι οποίοι εγκαταλείπουν πολύ μεγάλες ε, τράπεζες όπως η Goldman Sachs και αρχίζουν και εργάζονται σε κάποιες ε, μικρές επιχειρήσεις που όμως εξακολουθούν και διαχειρίζονται πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Είναι υπεύθυνε για πολύ σημαντικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να προβλέπονται παρεκκλήσεις για τις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα όσον αφορά τις ε, συναλλαγές των διαχειριστών. Οι διαχειριστές θα πρέπει να δημοσιεύουν τις συναλλαγές που κάνουν για οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ μέσα σε διάστημα δύο ημερών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον έχει προτείνει αυτό το ποσό των 20.000 ευρώ. Δεν προτείνεται κάποια αιτιολόγηση. Στο παρελθόν τα κράτη-μέλη είχαν την επιλογή να έχουν ένα όριο 5.000 ευρώ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχουμε περάσει τώρα στα 20.000 ευρώ, τα οποία δεν αποτελούν καν επιλογή αυτή τη στιγμή, αλλά επιβάλλονται ως υποχρέωση στην πρόταση οδηγίας. Επομένως, διέγραψα το σημείο αυτό, εφόσον δεν υπάρχει μια αιτιολόγηση ή κάποια μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως, οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να προτείνουν κάποιες άλλες απόψει για το σημείο αυτό. Εγώ πάντως δεν ήμουν απεπισμένο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα υποχρεωτικό μεσογειακό όριο 20.000 ευρώ. Μία από τις ε, σημαντικότερες συζητήσεις που είχαμε με τους ρυθμιστές και με τους ε, συναδέλφους ήταν ε, η διασυνοριακή επιτήρηση των δεδομένων που υπάρχουν στα βιβλία εντολών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ρυθμιστικές αρχές να καταφέρουν να δουν την κατάχρηση στις διασυνοριακές αυτές συναλλαγές οι εθνικές αρμόδιες αρχές επιτήρησης μας είπαν ότι πολλές φορές κάποιες συναλλαγές εμπλέκονται περισσότερο από 7 κράτη-μέλη, πολλές φορές και σε περιπτώσεις κατάχρησης της, αγορές, κατάχρηση της αγοράς. Δεν μπορούν λοιπόν να έχουν την απαραίτητη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται, προκειμένου να κάνουν μια αποτελεσματική επιτήρηση. Καθώς οι αγορές ολοκληρώνονται όλο και περισσότερο, ενοποιούνται όλο και περισσότερο, θα υπάρχουν όλο και υψηλότερε τάσει διασυνοριακής κατάχρησης της αγοράς. Θεώρησα λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων προκειμένου οι ε, εθνικές αρχές επιτήρησης να μπορούν να κάνουν την απαραίτητη επίβλεψη. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά, προτείνω η αρμόδια αρχή της πιο σχετικής επί της ουσίας αγοράς για μια συγκεκριμένη συναλλαγή θα πρέπει να έχει δεδομένα από όλα τα βιβλία των εντολών των ε, κρατών που έχουν συμμετάσχει σε μία συναλλαγή. Κατά αυτόν τον τρόπο η αρμόδια αρχή θα έχει τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να δει αν έχει γίνει κατάχρηση της αγοράς μέσω των βιβλίων εντολών. Στην έκθεση ε, Φέρμπερ αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στις, ε, στην επιτήρηση των συναλλαγών Θεώρησα πάντως ότι και στο δικό μου το κείμενο θα πρέπει να προβλέπετε μία πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα δεδομένα από όλα τα σχετικά βιβλία εντολών στα πλαίσια μιας συναλλαγής προκειμένου να υπάρχει αυτή η διασυνοριακή επίβλεψη. Ο άρθρο 48 και όπως λέγεται και μάλλον στην έκθεση Φέρμπερ φίτη στο σημείο 48 λέγεται ότι μπορούν να δίνονται πληροφορίες αυτές προς τρίτους. Ουσιαστικά συμπληρώνω εγώ αυτά τα οποία λέγονται στην ΜΥΦΗ, την Οδηγία για τις αγορέ Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να μπορεί να δημιουργηθεί η διαδικασία αυτή για τη συλλογή των δεδομένων από τα βιβλία των εντολών. Συνειδητοποιώ ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα πολύ σημαντικό ποσό πληροφοριών, για ένα πολύ σημαντικό όγκο πληροφοριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως να ξεκινήσει κάποια στιγμή η διαδικασία αυτή και να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια αυτής της διασυνοριακής ε, επίβλεψης των βιβλίων εντολών. Βρισκόμαστε σαφώς στην αρχή της όλης διαδικασίας. Πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια αρχή και να αρχίσουμε να εξετάζουμε αυτές τις πληροφορίες. η κυρία Πέτα Κάνεν και άλλοι κάναν κάποιες προτάσεις στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνε για τις ανταλλαγές των πληροφοριών θα πρέπει να κάνουν την επίβλεψη αυτή. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα εμπιστευτικότητα αυτή τη στιγμή. Πολλέ φορέ σε συνεργασία που έχουμε με τρίτε χώρε και ότι ενδεχομένω να μην έχουμε καταφέρει, ε, δεν θα καταφέρουμε να έχουμε εύκολα τι πληροφορίε αυτέ. Αν δείτε το άρθρο 17, δεν πρόκειται να σας διαβάσω, πάντως το άρθρο αυτό λέω ξεκάθαρα ότι ε, προβλέπεται μια νέα διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών όσον αφορά τα δεδομένα των βιβλίων εντολών. Πάλι όταν πήγαμε στη Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κόνγκ συλλέξαμε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για το τι μπορούμε να κάνουμε με, τις, με τα τιμολόγια τα οποία προτείνονται για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Δεν συζητήσαμε συγκεκριμένα για το ζήτημα αυτό με τον κύριο Φέρμπερ, πάντως και αυτό στην έκθεση ΜΥΦΙΤ έχει καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα όσον αφορά τα τέλη, όσον αφορά τις τιμές που επιβάλλονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ πέρα να αποφύγουμε καταχρηστικές πρακτικές από τους εμπλεκόμενους φορείς. Και γι' αυτό το λόγο λέμε εδώ πέρα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τέλος από τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αποφεύγεται ε, οποιοδήποτε φαινόμενο κατάχρησης αγοράς. Λέμε ότι πολλές φορές οι ψηλές τιμές ακύρωσης συνδέονται τελικά με καταχρηστικές πρακτικές. Αυτό το οποίο έκανα στην αρχή είναι να χρησιμοποιήσω ένα εφιστάμενο μοντέλο. Σε κάποιες συναλλαγές του Nasdaq είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται τα τέλη αυτά Σύμφωνα με το σύστημα Nasdaq, οι, οι άνθρωποι που συναλλάσσονται στα πλαίσια του Nasdaq θα πρέπει να καταβάλουν ένα ευρώ για συγκεκριμένε χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Επομένω, υπάρχει μια συγκεκριμένη, προτείνω μια συγκεκριμένη διάρθρωση των τιμών αυτών που θα πρέπει να υπάρχουν για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, Μπορούμε να δούμε πάντως μια γενικότερη τάση για την εισαγωγή των τελών αυτών, ακόμα και το Ιταλικό χρηματιστήριο και το Γερμανικό χρηματιστήριο προσπαθούν να εισάγουν παρόμοια τέλη. Υφίσταται η τάση αυτή, είναι μια πραγματικότητα και θα θυμάστε ότι όταν, συνεδριάσαμε στη Σιγκαπούρη και όταν έγινε μία συζήτηση για τις υπερβολικές τιμές εισαγωγής στο, χρηματιστήριο. Είπαμε τότε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, ένα συγκεκριμένο μοντέλο για την τιμολόγηση των συναλλαγών αυτών και δεν θα πρέπει οι φορείς να αποφασίζουν ανεξέλεγκτα για τις τιμές τις οποίες επιβάλλουν. Τώρα, όσον αφορά τους διαχειριστές, αν μπορούν να κάνουν μόνοι τους κάποιες ατομικές συναλλαγές για μια συγκεκριμένη περίοδο. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, είχαμε πει ότι θα έπρεπε να αποκλείσουμε τους managers από οποιαδήποτε συναλλαγή που κάνουν για δικό τους λογαριασμό. Θεωρήσω ότι αυτό ήταν κάπως υπερβολική προσέγγιση. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να δω αν μπορεί να υπάρχει ένα trading window, ένα παράθυρο συναλλαγής, δηλαδή μία χρονική περίοδος κατά την οποία θα μπορούσαν οι μάνατζερ να προχωρούν σε αυτές τις συναλλαγές. Προτιμώ να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση από να προχωρήσουμε σε μια συνολική απαγόρευση. Θα πρέπει και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών να δούμε πώς μπορούμε να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διαβολευτούμε και με τον κλάδο. Δεν είμαι υπέρ μιας απαγόρευσης. Πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες που να διευθετούν την αρχή και το τέλος της χρονικής αυτής περίοδου. Σε ορισμένε περιπτώσεις μπορούμε να πούμε ότι δεν θα επιτρέπεται συναλλαγή εκτός του παραθύρου συναλλαγής. Ξέρω ότι πολλές φορές οι μάνατζερ διαχειρίζονται μετοχέ της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Πρέπει λοιπόν και για τις σχετικές συναλλαγές να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Τώρα, όσον αφορά τις συναλλαγές υψηλή ε, συχνότητας. Όπω αναφέρεται και από την ΑΙΟΣΚΟ, τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Υποπτία Χρηματιστηρίων, ε, ε, δίνει τη δυνατότητα να εκτελούνται εντολέ σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και επομένω είναι πολύ πιο δύσκολη η ανείχνευση ε, του τι συμβαίνει. Αντί να μπούμε σε λεπτομέρειε στον κανονισμό αυτό για να πούμε τι πρέπει να κάνουμε, είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνουμε και ζήτησα να γίνει καλύτερη διερεύνηση για να αξιολόγησουμε τον αντίκτυπο των συναλλαγών υψηλή συχνότητα στη χειραγώγηση τη αγορά. Προτείνω λοιπόν να έχουμε μια συμβουλευτική επιτροπή Επιτροπή μέσα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, που θα πρέπει να υπάρχουν εθνικοί εμπειρογνώμονε για να εξετάσουν ε, τι συναλλαγέ υψηλή συχνότητα και τι ε, πιθανότητε χειραγώγηση τη αγορά. Θα έχουμε περισσότερε λοιπόν ε, γνώσει για, την... για τον τομέα αυτό για να ενημερωθεί κατάλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην, επιτροπή αυτή, στην έκθεση αυτή η Επιτροπή ε, απαγορεύει τρεις συγκεκριμένε καταχρηστικές πρακτικές, την παραποίηση δεδομένων, πρακτική συσσόρευση εντολών, ε, το quote stuffing, layering και spoofing δηλαδή προσπαθούμε να παραμείνουμε ενήμεροι όσον αφορά τις τάσεις ε, που ισχύουν σε αυτό το τομέα. Αυτό αντικατοπτρίζει και την τρέχουσα συζήτηση στις ε, ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Η Επιτροπή CFTC έχει δημιουργήσει την Επιτροπή TAC, που είναι μια συμβουλευτική επιτροπή για τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Επικεφαλής είναι ένας οικονομολόγος και υπάρχουν τέσσερις ομάδες εργασίας. Η πρώτη ασχολείται με τον ορισμό των συναλλαγών υψηλής συχνότητας. Η δεύτερη ομάδα εξετάζει το αν θα πρέπει να υπάρχουν πολλές κατηγορίες συναλλαγών υψηλής συχνότητας και συγκεκριμένα θα εξετάσει τις διακρίσεις ε, στις ε, ε, συναλλαγές που γίνονται κατά την είσοδο στην αγορά. Η τρίτη θα ασχολείται με την εποπτεία και την οικονομική ανάλυση για να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των συναλλαγών υψηλής συχνότητας σε σχέση με άλλες συχνότητες και η τέταρτη ομάδα εργασία θα ασχοληθεί με πιθανέ διαταραχέ στο εμπόριο από τι συναλλαγέ υψηλή συχνότητα. Αυτή η υποεπιτροπή στι ΗΠΑ θα καταλήξει σε κάποιε συστάσει και από τι συζητήσει που έχουμε κάνει με τι ΗΠΑ ε, ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ να μάθουν τι κάνουμε και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπάθησα λοιπόν και στην έκθεσή μου να το λάβω υπόψη μου αυτό, ιδίω όσον αφορά την κατάχρηση αγορά. Χαίρομαι που είδα ότι και ο κύριος Φέρμπερ στη ΜΥΦΙΝΤ ακολούθησε μια ισχυρή γραμμή για τα θέματα συναλλαγών υψηλής συχνότητας και νομίζω ότι η έκθεσή μου είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη και συμπληρώνει τη δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Φέρμπερ στη ΜΥΦΙΝΤ. Το επόμενο θέμα είναι η προστασία των ατόμων που καταγγέλουν παρατυπίες. Αν δείτε τα, τις τροπολογίες 45 47, τα άρθρα 28-29, ε, είναι νομίζω αυτονόητα. Προσπάθησαν να τα ενισχύσω. Εμπιστευτικότητα όλων των εμπλεκομένων για όλη τη διαδικασία. Τα άτομα που καταγγέλουν, χρειάζονται, που καταγγέλουν παρατυπίες χρειάζονται προστασία και στο χώρο εργασίας και υπάρχουν και εσωτερικοί μηχανισμοί οι οποίοι πρέπει να διοργανωθούν ε, εντός των επιχειρήσεων και αυτό είναι σύμφωνα με την οδηγία MIFID. Ε, υπάρχει παράλληλα και δυνατότητα να επανεξετάσουμε τα στοιχεία αυτά στο μέλλον, γιατί υπάρχουν ε, ταχύτατε εξελίξει ε, στην αγορά, ιδίω σε αυτέ τι συναλλαγέ. Θέλουμε λοιπόν διατάξει που να μπορούν να προσαρμόζονται στι μελλοντικέ εξελίξει. Γι' αυτό έχουμε πράξεις κατεξουσιοδότηση για να μπορούμε να ενημερώνουμε την νομοθεσία ανάλογα με τι καινοτομίε, στην τεχνολογία και στην κατάχρηση τη αγορά. Υπάρχουν και κάποιε άλλε πιο μικρέ αλλαγέ περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα, για να διευκρινίζονται ε, ε, γλωσσικά ε, ώστε να καλύπτονται όλες οι εξοχρηματιστηριακές συναλλαγές, να υπάρχουν αρκετοί πόροι για να καλύπτονται οι δραστηριότητες και να υπάρχει και αρμοδιότητα των καταλλήλων αρχών για να μπορεί να γίνεται η απαραίτητη έρευνα κάθε φορά. Θεώρησα ότι αυτά είναι σημαντικό να διευκρινιστούν. Αυτά περιλαμβάνονται στην πρότασή μου για τον κανονισμό. Ε, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα θέματα που εγώ παρέλειψα και θα θέλουν να προσθέσουν ε, οι συνάδελφοι και ευχαρίστω ε, θα κάνω και τη συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές στις προσεχέ εβδομάδες. Θεώρησα ότι είναι μια απλή οδηγία χρειάστηκαν 7 μήνε ε, για να οριστεί η συγητή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και αντί να ασχοληθεί με την ουσία της οδηγίας, ε, ασχολείται με τις διαδικασίες. Η κατάχρηση της αγοράς είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς αυξάνεται και αν δείτε ε, τα, τις οικονομικές ειδήσει, όλο και περισσότερο, περισσότερες περιπτώσεις κατάχρησης αγοράς αναφέρονται. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα μέσα και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τι αυξανόμενε περιπτώσει κατάχρηση τη αγορά. Εγώ προσπάθησα να περιοριστώ λοιπόν σε αυτήν την οδηγία σε, την τροποποίηση της θέσης σε ισχύ της οδηγίας για τις ποινικέ κυρώσεις, γιατί θα, πιστεύω ότι θα πρέπει να, να αρχίσει να ισχύει ένα χρόνο αργότερα και όχι δύο χρόνια αργότερα και είπε ότι θα πρέπει η ρήτρα αναθεώρησης να είναι στα δύο χρόνια και όχι στα τέσσερα χρόνια, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να εφαρμόζουν ποινικέ κυρώσεις για αυτό τον τομέα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δύο χρόνια αργότερα για να μπορούμε να κάνουμε τι απαραίτητε αλλαγέ ε, το συντομότερο δυνατόν για να μην περιμένουμε έξι χρόνια μέχρι να του δούμε αν λειτουργούν οι ποινικέ κυρώσει. Δεν έχω βάλει όμω πολλέ λεπτομέρειε σε αυτό το τομέα για να παραμείνει απλή αυτή η οδηγία σχετικά με τι ποινικέ κυρώσει. Ήθελα να το αφήσω στου εισηγητέ τη Επιτροπή Λίμπετο να μπουν σε λεπτομέρειε. Ε, αλλά ελπίζω να μην ε, σπαταλούν χρόνο για διαδικαστικά θέματα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αρλίν. Πολύ καλή έκθεση αυτή, νομίζω. Και ευχαριστούμε πολύ. Ε, σε ευχαριστώ εγώ για τη βοήθεια στους πολέμους επιτροπών, όπως τους αποκαλούμε. Και τον Ζων Πολ Γκοζέ, ευχαριστώ γιατί μας βοηθάει όσον αφορά τις επιτροπές. Περνούμε στους σκιώδεις εισηγητές, εκ μέρου του ΕΛΚ, ο Ζαν Πολ Γκοζές. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι εκτάκτος σήμερα. Ε, θα αντικαταστήσω το συνάδελφο που, τη συνάδελφο που υποχρεώθηκε να επιστρέψει στη Φινλανδία και θα προσπαθήσω με έξινο τρόπο να διαβάσω το σημείωμα που μου άφησε για να σας πω ποια είναι η άποψή της. Βέβαια, την κυρία Μακάρθη θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την πολύ καλή της εργασία και για τις τροπολογίες της και για τη μέθοδο εργασίας της, ώστε να έχουμε μια άριστη συνεργασία. Και την κυρία Μακάρθη θα ήθελα να τη συγχαρώ για τη διάθεσή της αυτή την ε, διαμεθοριακή, το διεθνικό έλεγχο να τον ενισχύσει και να δούμε αυτές τις αγορές που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα για μια επαγρύπνηση, για ένα έλεγχο και ταυτόχρονα όσοι δρούν στα πλαίσια αυτών των αγορών να έχουν ε, μια κατάλληλη επαγρύπνηση όπως πρέπει και αυτό είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Ε, αλλά στα πλαίσια που είναι τόσο περίπλοκα αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να συνεχιστεί. Λοιπόν, ε, και οι αρχές των κρατών μελών ε, ίσως δεν έχουν τα απαραίτητα κονδύλια για μια παρόμοια εποπτεία και μάλιστα αυστηρή. Γι' αυτό συνάδελφος θα ήθελε να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα αυτό για να έχουμε και συμπληρωματικά μέτρα για την κατάργηση ότι αυτή την κατηγορία αυτή εγκρίνεται αυτή η θέση και σε όσα λένε για μια κατηγορία ακριβώ θα ήταν ε, δύσκολα τα πράγματα και θα υπήρχαν ε, περισσότερες δυνατότητες καταχρήσεων. Ε, και η OTF ε, ακριβώς όπως έχει προταθεί από, για το MIFID από τον ε, κύριο Φέρμπερ αυτή η οδηγία για την αγορά χρωματοπιστωτικών μέσων και όλα αυτά που εφαρμόζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για όσους γνωρίζουν μυστικά θεωρείται ότι η παρόμοιοι κατάλογοι είναι κάτι το σημαντικό και αυτό και για να αποφύγουμε παρόμοιε καταχρήσει στην αγορά, αλλά για να υπάρξει εμπιστοσύνη στην αγορά. Άρα λοιπόν η ίδια θέση με εσά και επίση σα συγχαίρει για την πρότασή σα ώστε να συσταθεί μια επιτροπή συμβουλευτική πριν από τον Ιούλιο του 2014 για να δει τις ε, δυνάμει ε, χρήση αγορά και επίσης υποστηρίζει για μια βάση, την ιδέα για μια βάση διαπραγματεύσεων με κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να μην υπάρξουν καταχρηστικές εντολές διαχείρισης. Και αυτό το ποσό το οποίο αναφέρατε, 20.000 και κάτι, δεν είναι σίγουροι ότι είναι προς το συμφέρον της αγοράς να καταργηθεί το κατόφλι αυτό και μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κατόφλι χαμηλότερο ε, γενικό για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ρεαλιστική λύση. Και ακόμα ένα τελευταίο θέμα θα ήθελα να θίξει ορισμού του τι σημαίνει ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία σχετικά με αυτά τα παράγωγα, όσον αφορά αυτά, τα μέτρα όσον αφορά τις πρώτες γιατί θα πρέπει να δούμε τα δυνάμει προβλήματα όπως έχουν σήμερα για να έχουμε ένα πρακτικό ορισμό που θα μπορούσαμε να έχουμε μια προσαρμογή των όρων με τις συνθήκες όπως ισχύουν αυτές στην αγορά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ εξ ονόματος της ομάδας των Φιλεφέρων, Φιλίπ Πέκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος του κυρίου Κλίνς, ο οποίος ε, δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ και να διαβάσει την δήλωση αυτή την οποία μου έδωσε. Θα ήθελε καταρχάς να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία τα οποία θα ήθελε να θίξει. Καταρχάς, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, δεν συμφωνεί με τις τροπολογίες της ε, ε, εισηγήτριας που ουσιαστικά αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής της ε, οδηγίες αυτής στα ΟΤΕΕΦ, τους Εργανομένους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης. Όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες, είναι υπέρ των σχετικών τροπολογιών που θεωρούν ότι θα πρέπει να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών σε περίπτωση δημόσιας εξαγοράς. Όσον αφορά τους ε, καταλόγους εμπιστευτικών πληροφοριών, insiders lists, θα πρέπει πάλι εδώ πέρα να προβλέπονται κοινοί κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις οποιοδήποτε μεγέθους. Όσον αφορά το ποσό των 20.000 ευρώ, μπορεί να θεωρείται πολύ μικρό σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και υψηλό ποσό σε άλλα κρατημέλη. Θεωρεί λοιπόν ότι το σημείο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο στις περαιτέρω συζητήσεις που θα γίνουν. Επίσης είναι υπέρ του να υπάρχει ένα παράθυρο συναλλαγής, πρέπει όμως πολύ προσεκτικά να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του παραθύρου συναλλαγής. Όσον αφορά τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, Πιστεύει ο σκιωδησηγητής ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες αναλύσεις για να δούμε ποια είναι τα φαινόμενα κατάχρηση της αγοράς σε σχέση με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Θα πρέπει λοιπόν να συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμών για το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα την εποπτεία για το βιβλίο εντολών, θα πρέπει να υπάρχει όντως ένας μηχανισμός διασυνοριακός για την εποπτεία των βιβλίων εντολών, προκειμένου να αποφεύγονται τα, φαινόμενα, τα διασυνοριακά φαινόμενα κατάχρησης της αγοράς. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής ε, είναι υπέρ του όντως να δοθεί περισσότερο βάρος στη ρυθμιστική αυτή αρχή η οποία βρίσκεται στη χώρα όπου γίνονται σημαντικότερες συναλλαγές στα πλαίσια μιας ασυνοριακής ε, χρηματοπιστωτικής συναλλαγής. Ευχαριστώ πολύ εκ των Πρασίνων. Πασκάλ. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς από το ECR παρόν. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Πασκάλ. Ναι. Δεν θα σας πω τώρα όλη τη σειρά των σημείων με τα οποία σύμφωνα στην έκθεση αυτή, γιατί θα έτρωγε όλο το χρόνο μιλία μου. Γι' αυτό ακριβώ απλά και μόνο να υποστηρίξω ιδιαίτερα από πλευράς πρασίνων το σύνολο σχεδόν των προτάσεων που υποβάλλονται στην έκθεση αυτή για να βελτιώσουμε την εποπτεία της θέμα σχετικά με τις καταχρήσεις ε, σε παρόμοια θέματα και στα πλαίσια των όσων εμφανίζονται εδώ το πρώτο σημείο βλέπουμε είναι ότι το trading ε, το ιδιαίτερα συχνό και την πρόταση η οποία υποβάλλεται στην έκθεση από την συνάδελφο έχουμε ένα θέμα σχετικά με το ποσό που προτείνεται 250 εντολές για αυτές τις συναλλαγές ο αριθμός αυτός προέρχεται από μια ληφθής απόφαση στην, σε μια αμερικανική αγορά και στις συζητήσεις που είχαμε διάφορους που συμμετέχουν εκεί ε, άκουσα ότι θα μπορούσε κανείς να είναι περισσότερο φιλόδοξος για υψηλότερο αριθμό που είναι μια αυτορύθμιση ουσιαστικά της αμερικανικής αγοράς αυτός ο αριθμός 250 και γι' αυτό ακριβώς ε, θα μπορούσαμε και να το συζητήσουμε αυτό. Αν είναι ο κατάλληλος αριθμός συναλλαγών, μήπως θα μπορούσε να είναι υψηλότερος και θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, δεύτερο, για την εποπτεία αυτής της ε, καταχρήσης στα πλαίσια αυτής της αγοράς, ε, αυτός το cross-borders κλπ. Εδώ πρόκειται για σημαντικό στοιχείο. Βρισκόμαστε στην Ευρώπη και βλέπουμε με μια πολυδιάσπαση της αγοράς ε, και ο περίπλοκος αυτός χαρακτήρας ε, επιτρέπει χειραγωγή της αγοράς. Έτσι. Και νομίζω ότι το τίμημα είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να οδεύσουμε προς την κατεύθυνση που η συγγήτρια προτείνει να υπάρξει μια παγίωση των εντολών ώστε ρυθμιστές να μπορούν να έχουν μια συνολική εικόνα των θέσεων και των εντολών που δόθηκαν στις διάφορες πλατφόρμες. Και θα πρέπει να εργαστούμε και να δούμε πώς θα το πετύχουμε αυτό, αλλά επιμένω για την απόλυτη προτεραιότητα που θα πρέπει να αποδοθεί στο σημείο αυτό, σύμφωνα με την άποψη της ομάδος μας, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δούμε αυτές τις ε, καταχρήσεις αγοράς ε, της ε, χειραγωγής αγοράς. Και το τρίτο σημείο είναι οι κυρώσει. Εντάξει, διάφορα ρυθμιστικά μέτρα θα μπορούσαν να ισχύσουν, αλλά εάν δεν είναι στο κατάλληλα αντίστοιχη ποινή αυτό το πρόστιμο με τα κέρδη, τότε θα μπορούν πάντα να επιχειρούν να να χειραγωγήσουν την αγορά. Έτσι. Λοιπόν, σχετικά με την αρμόνιση αυτών των διοικητικών επίσης ποινών και κυρώσεων και να είναι αποτρεπτικός ο χαρακτήρας αυτών των ποινών γιατί σε ορισμένα κράτη, μέλη, ε, τα χρήματα που πληρώνει κανείς απρόστιμο είναι πολύ χαμηλό το ποσό και γι' αυτό ο καθένας μπορεί να προχωρήσει και θα χρειάζεται να δούμε... Ε, τις δέκα έτη που θα πρέπει να ισχύουν αυτές οι ποινές και άλλο είναι, άλλη είναι η ποινική διάσταση. Εδώ μιλάμε για διοικητικά μέτρα. Θα μπορεί κανείς να πετύχει μια εναρμόνιση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει την αποτελεσματικότητα αυτής της οδηγίας και να πετύχουμε μια καλύτερη ανιαγόρα. Ένα τελευταίο σημείο τώρα είναι ε, το πώς θα έχουμε τον συναγερμό, όπως τον αποκαλούμε, το καμπανάκι που θα χτυπάει εδώ που θα πρέπει να δούμε το, τα μέτρα που να ισχύουν για τις ε, ομάδες, για τις επιχειρήσεις, για τους ομίλους ε, και χρειάζονται μέτρα ώστε εκείνο που δίδει αυτό συναγερμό να ε, εκτός από την εσωτερική οργάνωση να υπάρξει και ένα κατάλληλο κύκλωμα που να πηγαίνει προς τα έξω από τη στιγμή που θα υπάρξει μια ένταση στην αγορά εσωτερικά. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία αλλά υπάρχει ένα σχετικά δυνάμεων και πιέσεις το ένα το άλλο. Λοιπόν, υπάρχει μια μέση επαφή με κάποιον τρίτο το ΕΣΜΑ, ας πούμε, αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ε, δηλαδή και σε εσωτερικό επίπεδο και προς τα έξω και έτσι θα μπορούσαμε κάπως να δείξουμε και <laughs> ανώνυμα τις πληροφορίες ε, και έτσι θα μπορούσαμε να καταστήσουμε αποτελεσματικό αυτοπιανισμό έτσι, σχετικά με το θέμα αυτό του συναγερμού της έγκαιρης προειδοποίηση ε, και ακόμα κάτι για μια ενδεχόμενη τροπολογία από εμά. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι συμφωνούμε ιδιαίτερα με όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αυτό το τελευταίο θα θέλαμε να θίξουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον από την ΚΟΕ παρόντα. Περνώ στον Godfrey Bloom. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, ε, γιατί ξέρω ότι έχετε καλές προθέσεις, αλλά μετά από πάνω από 30 χρόνια στο City του Λονδίνου, ξέρω ότι η αγορά καμιά φορά ε, είναι κατά του, του ρυθμιστή. Γιατί καμιά φορά οι ρυθμιστές νομίζουν ότι μέσα στην αλαζονία τους μπορούν να τα κάνουν όλα και φοβούμαι ότι και η Επιτροπή μπορεί να πέσει σε τέτοιο σφάλμα. Πριν από 12 χρόνια στο City ε, ήμουν στι οικονομικέ υπηρεσίε και προσπάθησαν οι Αμερικανοί να ρυθμίσουν αυτό το θέμα ε, με κάτι που αποκαλούσαν πράξη εξυγχρονισμού ε, των συναλλαγών. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Παρακαλώ να το εξετάσετε. Είναι ένα νόμο που πέρασε το 2000 στι ΗΠΑ. Και το αποτέλεσμα αυτού του νόμου ήταν ότι όλα βγήκαν εκτός ισολογισμού. Δεν άλλαξε τίποτα τελικά γιατί, ε, όπως σας είπα, τελικά η αγορά κερδίζει, η αγορά είναι ο νικητής. Υπήρχαν ε, ε, δυσμενείς επιπτώσεις ότι αντί να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, τα κάναμε χειρότερα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας προειδοποιήσω όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλοι ομιλητέ, ο Μάρκος Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με όλους εκείνους που επενούν την εισηγήτρια και την ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχει κάνει. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να προσέξουμε ε, να μην ε, μπερδέψουμε τις αρμοδιότητές μας. Εγώ δεν κάνω τίποτα για το δικό σας τομέα της κατάχρησης της αγοράς. Εγώ ασχολούμαι στην έκθεσή μου με την MIFID προσπαθώ να δω τι γίνεται στον τομέα της MIFID σχετικά με τα προϊόντα αυτά θα πρέπει αν αποφασιστούν αυτά τα οποία αποφασίζονται στη μύθη, να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και στην οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς. Το θέμα λοιπόν των οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης θα πρέπει να το συζητήσουμε για να υπάρχει συνέπεια και να μην έχουμε προβλήματα να μην ρυθμίζονται δηλαδή πράγματα ε, που πρέπει να ρυθμίζονται στη MIFID στην οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς. Ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει ε, να βάλουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό για την καταχρηστική καταχώρηση εντολής. Αυτό το 250 προς 1 ως λόγο εντολών προς συναλλαγές πρέπει να προσέξουμε πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε τη ρύθμιση αυτή μία φορά και όχι πολλές φορές. Να δούμε λοιπόν τι πρέπει να βάλουμε στη MIFID και τι πρέπει να βάλουμε στην οδηγία για την κατάχρηση των αγορών. Και πάλι για να ε, υπάρχει ε, συνέπεια μεταξύ ε, των αντιμετωπίσεών μας. Υπάρχει και έκθεσή μου για τη MIFID όπως γνωρίζετε και δεν θέλουμε να τα βάλουμε όλα ε, μέσα σε μία έκθεση. Δεν θέλουμε όλα να τα βάλουμε στον κόσμο της MIFID. Εσείς ενδεχομένως θέλετε να ελέγξετε και τη διασταυρούμενη χειραγώγηση αγοράς. Πρέπει να δούμε τι γραμμή θα ακολουθήσουμε, να δούμε ε, ε, ποια τακτική θα ακολουθήσουμε και το ίδιο να κάνουμε σε όλες τις οδηγίες. Ε, να προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε συνεπείς και χρονικά για να μην ε, ε, κάνουμε πράγματα που θα αποβούν εναντίον μας σε σχέση με τις αρμοδιότητές μας και του Συμβουλίου και αλλού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τόμας Μάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αλήν, άκουσες πολλά κομπλιμέντα και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να σε συγχαρώ για το έργο σου συνάδελφοι που ε, δουλεύουν στο City του Λονδίνου άκουσα που είπαν ότι ε, οι αγορές είναι πολύ έξυπνες. Ε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη στάση. Εγώ χαίρομαι που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση όπου μπορούμε να συζητήσουμε τις διάφορες απόψεις για να δούμε πώς να αντιμετωπίσουμε όλες τις λεπτομέρειες της αγοράς, γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να επέμβουμε στις αγορές. Θα πρέπει ε, να μπορούμε ε, να ελέγξουμε τις αγορές. Και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και για ε, τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Είναι τεράστια η κατάχρηση της αγοράς σε αυτό τον τομέα βάζοντας μια χρονική προθεσμία το 2015 νομίζω ότι είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Και όσον αφορά το θέμα του λόγου 250 προς 1, το ανέφερε και ο Πασκάλ, να προσέξουμε να μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, αλλά λαμβάνοντα υπόψη και αυτά που συμβαίνουν και στην Αμερικανική αγορά, νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε μια λογική στάση. Έχω και μια ερώτηση στην τροπολογία 26 σχετικά με τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων σε αγορά ανάπτυξης. Γιατί διαγράφεται αυτή η παράγραφος, δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους μεγάλους επενδυτές, ε, αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια αγορά, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο προσώπων ε, ώστε να μας δίνει, να δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ένα κατάλογο με περιγραφή των ατόμων που έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Το βρίσκω σκόπιμο αυτό. Κάποια λύση πρέπει να βρούμε. Με ενδιαφέρει λοιπόν γιατί το έχεις, προτείνει να διαγραφεί αυτή η παράγραφος. Άλλο ένα σημείο για τις κυρώσεις που υπάρχουν και πόσο αποτρεπτικά πρέπει να δρουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κυρώσεις. Χρειαζόμαστε θεσμικά όργανα, χρειαζόμαστε διαρθρώσεις. Τα κράτη-μέλη πρέπει να παίζουν ένα πιο ενεργό ρόλο από ό,τι μέχρι τώρα. Και Πιστεύω ότι ε, το σημαντικό είναι ότι ε, η διασταυρούμενη χειραγώγηση αγοράς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι πρόθεσή μας να το κάνουμε. Και ο Μάρκους Φέρμπερ θα φροντίσει ώστε να έχουμε τελικά δύο εκθέσεις ε, για δύο οδηγίες που να μην είναι αντιφατικές αλλά να αλληλοσυμπληρώνονται και την επόμενη φορά ε, νομίζω ότι θα μπορούμε ε, να έχουμε στοιχεία και για ε, τη διαβούλευση στον κλάδο, για να ξέρουμε τι συμβαίνει στην αγορά, τι συμβαίνει στον επαγγελματικό χώρο. Και πιστεύω ότι όταν ε, προτείνουμε λογικές ρυθμίσεις της αγοράς δεν είναι κάτι υπερβολικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας να κάνω το ακόλουθο σχόλιο. Ξέρετε ότι περισσότερες συνεδριάσεις ε, μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου εκτός από τις συνεδριάσεις που γίνονται στο Στρασβούργο. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλος το λόγο αυτή τη στιγμή. Επομένως, θα ήθελα να κάνω αυθόρμητα κάποιες παρατηρήσεις. Όπως μας είπε και η Αρλίνα, όντως είχαμε μια πολύ επικοδομητική επίσκεψη της Επιτροπής μας στην Ασία, όπου είμαστε σε θέση να έρθουμε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και να θέσουμε πολλές ερωτήσεις. Πρέπει όμως να πούμε ότι όντως οι αγορές τους δεν είναι τόσο πολύπλοκες και ότι δεν καλύπτουν τόσα πολλά στοιχεία διαπραγμάτευσης όπως για παράδειγμα οι αγορές του Λονδίνου. Ωστόσο ήταν πολύ επικοδομητική η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στην Ασία και βλέπουμε ότι η Αρλίν έχει συμπεριλάβει στο κείμενό τη ένα μεγάλο μέρο από τα στοιχεία αυτά τα οποία συζητήσαμε στην Ασία. Όσον αφορά τα OTF τώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο τα καλύψαμε και στην έκθεση του Μάρκου Φέμπερ για το MIFID. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω πώ μπορούμε να εντάξουμε τελικά την κατηγορία αυτή και ενδεχομένω εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Αναρωτιέμαι αν είναι σωστό να έχουμε μία απαγόρευση των σχετικών κεφαλαίων, δηλαδή να μην μπορούμε να αναφερθούμε στα κεφάλαια αυτά στα πλαίσια των οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε την κατηγορία του market making capital χωρίς να χρησιμοποιούμε πολλούς διαφορετικούς μαθηματικούς ε, τύπους. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε απλώς ένα ποσοστό. Ενδεχομένως ε, ένα μικρό ποσοστό τέτοιων κεφαλαίων να μην ε, προκαλεί κάποιο πρόβλημα, αρκεί το ποσοστό να είναι χαμηλό. Αυτή είναι μια πρώτη ιδέα την οποία είχα, ζήτημα το οποίο άπτε περισσότερο του αντικειμένου της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Σε μια τέτοια όμω περίπτωση, εφόσον επιτρέψει το μικρό ποσοστό, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν υπάρχει και μια κύρωση, αν υπερβεί κάποιο το ποσοστό αυτό. Επίσης, Είπαμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει ε, η νομοθεσία που υπάρχει για την καταπολέμηση τη κατάχρηση τη αγορά δεν ευνοεί κάποιε μακροπρόθεσμε επενδύσει. Επομένως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες διαφορετικές κατηγορίες εμπιστευτικών πληροφοριών. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας τέτοια προσέγγισης, αλλά θα μπορούσαμε και αυτή να την εξετάσουμε. γιατί ξέρετε ότι είμαστε σαφώς υπέρ των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις αυτές. Διαβάζοντας λοιπόν το σχετικό άρθρο, άρχισα να ρωτιέμαι για το ποια προσέγγιση θα πρέπει να εγκρίνουμε. Είμαι υπέρ του να υπάρχει μια εποπτεία όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές ε, συναλλαγές και όσον αφορά τη διασυνοριακή εποπτεία των βιβλίων εντολών. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα πρότυπα και να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τον ίδιο τρόπο τα βιβλία εντολών από τη μία χώρα στην άλλη. Σε μία σχετική αιτιολογική σκέψη του κειμένου και στην ε, ΜΥΦΙΤ έχουμε αρχίσει να ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε έναν πολύ καλύτερο εποπτικό έλεγχο στο μέλλον ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξο, πρέπει πάντως έστω και τώρα να θέσουμε τη βάση και σε αυτή τη νομοθεσία και στις υπόλοιπες σχετικές νομοθεσίες που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Τώρα όσον αφορά την βάση τέλους που χρησιμοποιείται, όσον αφορά τις εντολές. Πάλι εδώ θεωρώ ότι η ιδέα που έχει προταθεί είναι πολύ καλή και όπως μας είπε και η Αρλίν, έχει δοκιμαστεί ήδη σε διάφορες κατηγορίες συναλλαγών. Δεν ξέρω αν θα πρέπει το τέλος που προβλέπεται να είναι ανεντολή ή αναμήνυμα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει κάποια διαφορά. Σε ορισμένε περιπτώσεις, ακόμα και με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, το γεγονός ότι καταχωρούνται συγκεκριμένες εντολές, είναι συγκεκριμένο αριθμός εντολών, δεν απαραίτητα κάτι το αρνητικό. Σε ορισμένε περιπτώσεις υπάρχουν μηχανισμοί που αποκλείουν τις πιο ακραίες τιμές. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα, αν το τέλος θα πρέπει να υφίσταται ανά εντολή ή ανά μήνυμα. Ξέρετε ότι το τέλος κάθε φορά υπολογίζεται μια συγκεκριμένη, με ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Πολλές φορές οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μας λένε ότι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας χρησιμοποιούν ένα μεγάλο ποσοστό της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής που προβλέπεται για τον καθορισμό του τέλους. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και στα πλαίσια του MIFID, αλλά καθότι τίθηκε το ζήτημα εδώ πέρα, πιστεύω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό από το συγκεκριμένο κείμενο για την καταπολέμηση κατάχρηση αγορά. Σίγουρα θα πρέπει να διευθετηθεί στα πλαίσια τη MIFID. Όσον αφορά τώρα την οδηγία, όντως να γνωρίσουμε ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι η πλέον αρμόδια προκειμένου να αποφασίσει για τις ποινικέ κυρώσεις που θα πρέπει να προβλέπονται. Και ότι θέλουμε τελικά να έχουμε ποινικέ κυρώσεις και δεν θα πρέπει αυτό βέβαια να επηρεάζεται από το αν το ζήτημα αυτό εξετάζεται από τη δική μας την Επιτροπή ή από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ή ακόμα και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν νομίζω πάντως ότι θα πρέπει αποσπασματικά κάθε φορά να αποφασίζουμε για αυτές τις ποινικέ κυρώσει και κατά περίπτωση τελικά να βλέπουμε ποιες θα είναι οι κυρώσει που θα πρέπει να ισχύουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που να ισχύουν σε κάθε περίπτωση και που να τηρούνται από όλου. Θα θέλαμε λοιπόν στη δική μας την Επιτροπή να έχουμε κάποιες ε, βασικές αρχές όσον αφορά τον καθορισμό των ποινικών κυρώσεων. Είναι πολύ σημαντικό να μην καταλήξουμε όμως σε μία μέγιστη εναρμόνιση, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και αυτό γιατί υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία ήδη προβλέπουν πάρα πολύ αυστηρέ ποινικέ κυρώσει σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη που έχουν πιο ήπιε και σε σχέση με άλλα που δεν έχουν καθόλου ποινικέ κυρώσει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια ελάχιστη εναρμόνιση, όπως, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν λάθος πάντως να υπάρξει μία σύγχυση να υπάρχουν ε, μεταξύ διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Άλλο πράγμα είναι οι διοικητικές κυρώσεις και άλλο πράγμα οι ποινικές κυρώσεις. Για μια συγκεκριμένη κατάχρηση τη αγορά θα μπορούν να προβλέπονται και διοικητικέ κυρώσει και εφόσον κριθεί αναγκαίο, αλλά ακόμα και ποινικέ κυρώσει. Στην ε, οδηγία για την ε, χρήση των κεφαλαίων κάνουμε μία αναφορά και σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι οι ποινικέ κυρώσεις και οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να συνεπάρχουν. Έχει ασχοληθεί πάντως και η Αρλίν με το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα εξετάσει και αυτή το ζήτημα αυτό στα πλαίσια του CRD. Αυτά είχα να σας πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρλίν για την ε, ιδιαίτερα καλή και διαφωτιστική αυτή της έκθεση. Μπορούμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον το θέλει η συγγήτρια. Νομίζω ότι είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπροσωπείτε. Έχετε το λόγο λοιπόν. Like to thank... Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Αρλίν Μακάρθη για την έκθεση που μας παρουσίασε είναι προς την ίδια κατεύθυνση όπως και η γραμμή της Επιτροπής όσον αφορά την ε, βελτίωση του καθεστώτος ε, της αγοράς. Υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία στα οποία προτιμούμε να κρατήσουμε το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής γιατί θεωρούμε ότι είναι αναλογικά όσον αφορά την εξαίρεση για τον κατάλογο αυτών ε, που μεταφέρουν εμπιστευτικέ πληροφορίε, Νομίζω ότι ήταν πολύ συγκεκριμένο μέτρο και ισορροπημένο. Θέλω να τονίσω, όπως ανέφερε και η ίδια η συγγήτρια και ο κύριος Φέρμπερ, ότι πρέπει να παραμείνει η συνέπεια και η συνοχή μεταξύ των δύο θεμάτων. Κάποια από τα στοιχεία αυτής της έκθεσης ίσως στο νομικό πλαίσιο ταιριάζει καλύτερα στη MIFID. Όλα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εκτός από το σημείο της ε, αφαίρεσης της κατηγορίας OTF. Αν όμως αποφασιστεί ότι ε, αφαιρείται η κατηγορία OTF των οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης, ε, είναι σαφές ότι οποιοδήποτε είδος διαπραγμάτευσης από πλατφόρμες θα πρέπει να καλύπτεται από την οδηγία για την κατάχρηση αγοράς. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή η ΕΣΜΕ, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ασχολείται με θέματα συναλλαγών υψηλής συχνότητας και υπό το πλαίσιο της κατάχρησης της αγοράς και υπό το πλαίσιο της MIFID. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η δουλειά και είναι σημαντικό να συνεχιστεί. Και για τις κυρώσεις θέλω να αναφέρω ότι και εδώ πρέπει να τηρήσουμε μια συνεπή προσέγγιση με αυτά τα οποία συζητούνται σε άλλες προτάσεις, όπως η οδηγία για τα, την κεφαλαιακή επάρκεια, για την ΟΚΑ 4 και για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και το χρονικό πλαίσιο που δίδεται για την εφαρμογή των μέτρων στα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι επαρκές για να είναι σωστό το τελικό νομοθετικό αποτέλεσμα. Το συμπέρασμά μου τελικά είναι ότι το Κοινοβούλιο βρίσκεται στη σωστή πορεία για το θέμα αυτό και προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συζήτηση. Ο σκοπός είναι οι συνομοθέτες να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του, της τελευταίας διάσκεψης κορυφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ξαναδίνω το λόγο στην Αρλίν. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί είπα από την αρχή ότι δεν ε, έχω κάποια τελικά διαμορφωμένη στενή άποψη για θέματα λεπτομέρεια. Είμαι ανοιχτή και θα περιμένω τις απόψεις σας για να διαμορφώσουμε καλύτερα αυτή την έκθεση. Για το αν υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ αυτού του κανονισμού για την κατάχρηση αγορά και τη MIFID, θα ήθελα να πω ότι καθόλου δεν τίθεται έτσι το θέμα και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Φέρμπερ να σεβαστείτε ότι όταν εγώ ασχολούμαι με ένα κανονισμό ή οδηγία ε, ε, όπου υπάρχει ε, συνεχώς αυξανόμενη κατάχρηση αγοράς και όπου υπάρχει όπου αναφέρεται ότι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας ε, είναι κάτι που συνεχώς ε, δημιουργούν αυξανόμενη κατάχρηση αγοράς είμαι υποχρεωμένη να το αναφέρω αυτό είμαι υποχρεωμένη να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι σημαντικό θέμα ε, για την κατάχρηση της αγοράς. Ε, είναι τομέας όπου η κατάχρηση της αγοράς αυξάνεται, άρα κάπου πρέπει να το αναφέρουμε. Λόγω του χρονοδιαγράμματος, λόγω του πιεσμένου χρονικού πλαισίου, δεν είχα το χρόνο να δω τι ακριβώς υπάρχει μέσα στη MIFID. Πιστεύω ότι όταν μας λένε οι ρυθμιστικές αρχές ότι το να δημιουργείται μεγαλύτερος κατακαιρματισμός ε, δυσκολεύει περισσότερο την ανείχνευση της κατάχρησης αγοράς και τη δίωξή της, είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρω στην εκθεσή μου. Το έχουν πει οι ρυθμιστικές αρχές, αλλά πρέπει και εγώ στην εκθεσή μου να το αναφέρω. Όπως είπα, υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία ακόμη χρειαζόμαστε πολλή δουλειά και ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας και θα χαρώ πολύ αν έρθουν οι συνάδελφοι και μου προτείνουν κάτι στους τομείς αυτούς. Όσον αφορά την απάντηση της Επιτροπής ε, για την παρέκκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλετε να το κρατήσετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέλω να πω στην Επιτροπή, δεν το ζήτησαν καν αυτό. Το βλέπουν από μόνες τους ότι ε, ως ε, σημαντικό κομμάτι της οδηγίας αυτό υπάρχει και θέλουν να συμμορφωθούν προς αυτό. Εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να θέλετε να το κρατήσετε. Θέλετε να βρείτε έναν τρόπο να ελαφρύνετε το διοικητικό φόρτο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσετε αυτή τη διοικητική ελάφρυνση όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν λένε ότι χρειάζονται κάτι τέτοιο. Δεν είναι και πολύ σημαντικό το να κρατήσετε ένα κατάλογο με τα άτομα που χειρίζονται εμπιστευτικέ πληροφορίε. Μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αφού δεν το έχουν ζητήσει δεν χρειάζεται να το προσφέρετε δεν έχει ξεκινήσει ε, συζήτηση από αυτού. Το μόνο που έχει ξεκινήσει είναι μια συζήτηση που λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε από αυτού και έχει ε, ζητηθεί μεγαλύτερη έρευνα για το τι πρέπει να κάνουμε. Με κάθε σεβασμό προς την Επιτροπή πιστεύω ότι εμείς πρέπει να θέσουμε ε, τους όρους ως εκλεγμένο όργανο και θα πρέπει να ζητήσουμε από την ΕΣΜΑ να μας πει τι κάνει σε αυτό τον τομέα δεν πρέπει να περιμένουμε απλώ να δούμε τι θα βγάλει τελικά η ΕΣΜΑ, αλλά πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ότι ε, θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Όπω και άλλα θεσμικά όργανα σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Και εμένα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα κατάχρηση τη αγορά, όχι τα άλλα θέματα τα οποία προφανώ θα τα ρυθμίσει η MIFID. Ο Πασκάλ ανέφερε το θέμα των διοικητικών κυρώσεων. Είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερέστερα, νομίζω και η πρόεδρος ε, το ανέφερε, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα και την ισχύ των διοικητικών κυρώσεων. Δεν μιλάμε για κλήσεις της τροχέας. Είναι πολύ συγκεκριμένα εργαλεία που πρέπει να έχουν αποτρεπτικό ρόλο για την κατάχρηση της αγοράς και ευχαρίστω λοιπόν να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ τον κύριο Γκοζές για τα σχόλια που έκανε εκ μέρους της κυρίας Πετκάνεν. Διμερώς το έχουμε συζητήσει μαζί της ε, πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο. Ευχαριστώ και τον κύριο Μαν για τα σχόλιά του. Είναι το πρώτο σχέδιο της έκθεσης αυτής και θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Ξέρω ότι πρέπει να το επεξεργαστώ περισσότερο. και όσοι έχουν εμπειρία επί του θέματο, καλό θα ήταν να με βοηθήσουν. Και περνώ στον κύριο Μπλουμ. Εγώ ξέρω ότι ο κύριο Μπλουμ πολλέ φορέ παρεμβαίνει ε, και προσπαθεί να, να μου κάνει κήρυγμα. 35 χρόνια στο City του Λονδίνου. Φαντάζομαι ότι είστε απόλυτα αμερόληπτος για το τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον κανονισμό. Ε, είπατε ότι πριν από 12 χρόνια ήσασταν στην αγορά. 12 ε, χρόνια είναι μεγάλο διάστημα. Είσαστε πολύ μακριά από τι αγορέ γιατί αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Και θα προτιμούσα να έχω τη δική μου άποψη το τι κάνουν οι ρυθμιστικές αρχές, γιατί εγώ καθημερινά τους παρακολουθώ. Ξέρουμε ότι πολλές επιχειρήσεις, κακές επιχειρήσεις προσπαθούν να παρακάψουν τους κανόνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θεσπίζουμε κανόνες. Ευχαρίστως λοιπόν ό,τι επικοδομητικά σχόλια έχετε κύριε Μπλουμ να τα λάβω υπόψη. Αλλά όταν έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά οικονομικών υπηρεσιών θα έχουμε και διασυνοριακές ε, συναλλαγές αλλά πρέπει να έχουμε και κανόνες διασυνοριακούς. Αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα κράτος, σημαίνει περισσότερη Ευρώπη και φαντάζομαι ότι πρέπει να το δεχτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 8η Μαΐου. Θα τις εξετάσουμε τις τροπολογίες αυτές στη συνέχεια Α, Μάρκου, συγγνώμη, θέλει το λόγο, δεν Μία ερώτηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Για να είμαστε συνεπείς, ε, πράγμα το οποίο όλοι θέλουμε. Για τη δική μου έκθεση, νομίζω η συζήτηση είναι τέλη του μηνός μετά από την εβδομάδα του Στρασβούργου. Και όσον αφορά τις ψηφοφορίες, νομίζω κάπως πρέπει να συνεννοηθούμε θα ήταν επικίνδυνο να ε, έχουμε την ψηφοφορία πρώτα για το ένα και μετά για το άλλο. Κάπως μαζί πρέπει να τα συγχρονίσουμε. Πρέπει να συντονιστούμε κάπως. Κύριε Μακάρθη. Απολύτως συμφωνώ μαζί σας. Ναι, ναι. Θα φροντίσουμε και οι δύο εκθέσεις να συζητηθούν, να ψηφιστούν μαζί. Μάλιστα, θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. Θεωρητικά η ψηφοφορία θα γίνει στις 9 ε, Ιουλίου. Άρα πετυχαίνουμε αυτόν τον συγχρονισμό. Αν γίνουν βέβαια αλλαγέ ε, για τη μία έκθεση, θα έχουμε αλλαγέ και στην άλλη. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε συντονισμένα και για τα δύο ζητήματα. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Άρα θεωρητικά Πηγαίνουμε μάλλον για, τον, για την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Και κατά αυτόν τον τρόπο παραμένουμε συντονισμένοι με την ΜΥΦΙΔ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι όλοι έτοιμοι για το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 5, ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Βλέπω ότι η συγγήτρια είναι εδώ. Βλέπω επίσης και τον εκπρόσωπο από την ομάδα των σοσιαλιστών. Ο Σβέν θα έρθει από τους Πρασίνους. Οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων δεν γνωρίζετε. Νομίζω ότι θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο προτού φτάσουμε στις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Πρέπει να εξετάσουμε στις 11.30. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε να περάσουμε ευθύ αμέσω στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης ελκυστικό των επενδύσεων στην Ευρώπη. Αν είστε έτοιμοι ρόδι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή ε, «Επενδύομαι στην Ευρώπη» ε, πραγματεύεται ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζουμε για πρώτη φορά. Οι επενδύσεις είναι στην καρδιά πολλών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών θεμάτων και παρενέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να προωθήσουν τις επενδύσεις. Ε, πήρα αυτή την πρωτοβουλία για την έκθεση και ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να την εκπονήσω ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και στο διεθνές ε, στερέωμα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για να δώσουμε μια όθηση στις επενδύσεις μας. Η έκθεση παρουσιάζει καταρχάς το περιβάλλον το διεθνές. Βλέπουμε ότι η ανάκαμψη έρχεται αργά και είναι πολύ ευαίσθητη. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αφενός να είναι παρούσα στη διεθνή σκηνή και να συμβάλλει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη ε, ενδυνάμωση του διεθνούς εμπορίου ε, και των ανοιχτών συνόρων και αφετέρου θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει ένα περιβάλλον ανάπτυξης ε, διεθνές το οποίο ελπίζουμε ότι θα έλθει ε, σύντομα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς πρέπει να δει ποια είναι τα, τα πλεονεκτήματά της αφενός η ζώνη ευρώ, η σταθεροποίηση της ζώνης ευρώ είναι ένας πρώτος στόχος διότι αποτελεί ένα μεγάλο ατού τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις εξωτερικές επενδύσεις. Ε, απ' την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσουμε τη θέση της πρώτης ε, ε, αγοράς επενδύσεων που είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να μην αφήσουμε να χάνουμε έδαφος από άλλες αναδυόμενες δυνάμεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα. Είπαμε αφενός η αστάθεια στη ζώνη ευρώ είναι μεγάλο μειονέκτημα για εγχώριες και ξένες επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πώς θα σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα ευνοήσει την ρευστότητα προς την ε, πραγματική αγορά ε, και πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα διαφορετικά μας προβλήματα. Διότι για να προωθήσουμε τις επενδύσεις πρέπει να δούμε όχι τις επενδύσεις μόνο ως μέσο όρο ευρωπαϊκό, αλλά να δούμε οι επενδύσεις πώς κατανέμονται και στις διάφορες ε, ε, χώρες μέλη και πώς οι επενδύσεις ε, μπορούν να προωθηθούν από τις διάφορες περιοχές. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό ότι έχει κάνει στην έκθεσή μας γνωμοδότηση και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία έχει ενδιαφέρουσες ιδέες να μας δώσει σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει παράλληλα με τα πλεονεκτήματά μας να δούμε πώς θα λειτουργήσει και η εσωτερική αγορά. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα δώσει μεγάλες ευκαιρίες νέες επενδυτικές ευκαιρίες, η απελευθέρωση πολλών επαγγελμάτων, η ενδυνάμωση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων θα δώσει ευκαιρίες ανάπτυξης των υπαρχουσών ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη, θα έλξει ξένες επιχειρήσεις, διότι θα δημιουργήσει μια μεγάλη αγορά και δεύτερον θα δώσει νέες ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις με το άνοιγμα των ε, διαφόρων επαγγελμάτων. Ε, παράλληλα η Ευρώπη πρέπει να δούμε πώ θα αξιοποιήσει τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατή, παραδείγματο χάρη το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό πώ θα το κρατήσει ε, ενημερωμένο και προσαρμοσμένο και ανταγωνιστικό στι νέε εξελίξει. Εκεί η παιδεία μα και η επαγγελματική ενασχόληση, ε, επαγγελματική επιμόρφωση έχει πολλά να προσφέρει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η παιδεία ε, μπορεί να είναι και ένας χώρος επενδύσεων, όχι μόνο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και επενδύσεων νέων επιχειρήσεων ε, ή κοινών επιχειρήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η Μεγάλη Βρετανία, κυρία Πρόεδρε, αποτελεί ένα παράδειγμα προς αυτό το τομέα αξιοποίησης του χώρου της παιδείας για ανάπτυξη επενδύσεων. Ε, λοιπόν νομίζω ότι η Ευρώπη με την ε, φήμη την διεθνή που έχει πρέπει να αξιοποιήσει και το χώρο της παιδείας για να έλξει επενδύσει στον τομέα αυτό. Απ' την άλλη πλευρά το επίπεδο ζωής ε, στην Ευρώπη ε, η, με ό,τι σημαίνει αυτό, κοινωνικές προστασίες, πολιτισμική ζωή είναι στοιχεία σημαντικά για την έλξη ξένων επενδυτών. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, η έρευνα και η καινοτομία χαρακτηριστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού πνεύματος πρέπει να μπουν πιο πολύ στην πολιτική μας κάτι το έχει τονίσει η επιτροπή μας πολλές φορές στην πολιτική μας τόσο για την ε, ε, παραγωγή έρευνας όσο και για την αξιοποίησή της και την διάθεσή της από τις επιχειρήσεις ε, είναι πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε το ρόλο των διαφορετικών ταμείων. Αυτό θα το τονίσει στη γνωμοδότησή της και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει ακόμη μια φορά, δίνει έμφαση και η έκθεση εκεί, ότι τα διαφορετικά ταμεία στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, μην ξεχνάμε ότι είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης των σχεδίων μας. Και πρέπει όλα αυτά και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο να το εντάξουμε. Απ' την άλλη πλευρά η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις ε, ελεύθερες ε, ζώνες συναλλαγών, να προωθεί τις ελεύθερες ζώνες συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί αυτό θα δώσει ζωντάνια ε, στις δικές μας επενδυτικές, εμπορικές και επενδυτικές ικανότητες. Και επίσης η ε, η αμοιβαιότητα με ε, της πρόσβασης σε δημόσιες ε, αγορές όπως είναι ε, αυτό το οποίο προωθεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει με νέες δυνατότητες τόσο στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρεθούν στη διεθνή σκηνή όσο και καλύτερους, διαφανέστερους και ισότιμους όρους στις ε, μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές ε, εταιρείε να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία αποτελούν θέματα που τα έχουμε αναφέρει με την ευκαιρία ε, διάφορων εκθέσεων και ε, resolutions από την Επιτροπή μας θα πρέπει να τα εντάξουμε σε ένα συνεκτικό σχέδιο. Γι' αυτό η έκθεση τονίζει ότι αφενός πρέπει τα κράτη-μέλη με τη Eurostat να συνεργαστούν ούτως ώστε να έχουμε ειδικού δείκτες για τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος στις επενδύσεις. Πρέπει να στοχεύσουμε δηλαδή πιο συγκεκριμένα στο πώς θα αναδειχθεί η ανάγκη και η πρόοδος δημιουργίας επενδυτικού ε, πνεύματος. Απ' την άλλη πλευρά, στην προσπάθεια 2020, μεταξύ των ε, φάρων, των προγραμμάτων φάρων μας, πρέπει να είναι ε, και η επενδυτική προσπάθεια. Πρέπει να γίνει σαφής και να μην χαθεί σε γενικότερα πλαίσια. Γι' αυτό το λόγο ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει μια ε, communication μέσα στην οποία θα βλέπουμε πώς η Ευρώπη προχωρεί προς την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της, την αντιμετώπιση των αδυναμιών της ε, για να προωθεί τις επενδύσεις εγχώριες και ξένες γίνεται σαφής η αναφορά και η διαφορά μεταξύ εγχωρίων και ξένων επενδύσεων στην έκθεση και πώς θα προχωρήσει σε ε, προτάσεις στρατηγικών και νομοθετικών προτάσεων όπου χρειάζεται για να δημιουργηθεί αυτό το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον. Ε, πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσουμε και σε ένα παρατηρητήριο επενδύσεων, επενδυτικής προσπάθειας στην Ευρώπη, διότι ε, δεν είναι μόνο να δούμε σε πλαίσιο γενικό πώς προωθείται η επενδυτική δραστηριότητα στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε πώς κατανέμεται και στο πλαίσιο των κρατών μελών, διότι θα πρέπει να δούμε καλύτερα πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας, κράτη-μέλη, περιφέρειες, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε συγκριτικά και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα που έχουν διάφορες περιφέρειες, διάφοροι επενδυτικοί τομείς για να δημιουργήσουμε μια περισσότερο συνεκτική και αποτελεσματική ε, επενδυτική προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτά είναι σε γενικές γραμμές, ε, ε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προτάσεις της της έκθεσής μας επαναλαμβάνω είναι ανάγκη να βρεθούμε σε ένα πλαίσιο συνεκτικό στρατηγικό και να έχουμε εργαλεία παρατήρησης και παρακολούθησης της προσπάθειας. Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση. Περνάω στην ομάδα των σοσιαλδημοκρατών Μόιχα Κλέβερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της πολιτικής μου ομάδας ακούμε πάρα πολλά πράγματα για την ε, ανάγκη που υπάρχει για μεγαλύτερες επενδύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτή για μια έκθεση για την ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Μια έκθεση λοιπόν που παρουσιάζεται στην ε, Επιτροπή μας και που ουσιαστικά θα έπρεπε μέσω αυτής να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις ε, δυνατότητες ελκυστικότητας επενδύσεων στην Ευρώπη. Όπως λέγεται και στην έκθεση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε δύο συγκεκριμένους δρόμους. Από τη μια της δυνατότητας, τη δυνατότητα ανάπτυξη περαιτέρων επενδύσεων και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του παγώματος κάποιων επενδύσεων επιτόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να δούμε τη θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές πολιτικές, τις πολιτικές επενδύσεων ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε την πολιτική συνοχή, καθώς επίσης και τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική συνοχή εξυπηρετεί τις ανάγκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να τροποποιήσει τους κανονισμούς όσον αφορά την πολιτική συνοχής για τα επόμενα έτη και όντω είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι δαπάνε που προέρχονται από την πολιτική συνοχή προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποιε επιπτώσει από την κρίση στι πόλει, στι περιφέρειε, σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο μπορεί η πολιτική συνοχή τελικά να προωθήσει και τι επενδύσει στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίση να πω ότι τα διαφορετικά ταμεία μπορούν να έχουν ένα καταλητικό ρόλο προκειμένου να προσελκύσουν νέε επενδύσει και να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο μόχλευση στα πλαίσια του προπολογισμού προκειμένου να δημιουργηθούν και περαιτέρω επενδύσει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε όλους τους τομείς τα οποία μπορούν να έχουν ε, ένα πολλαπλασιαστικό φαινόμενο στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού. Προπολογισμού, με συγχωρείτε, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ε, νέα μέσα χρηματοδότησης... προκειμένου να γίνουν ε, αηφόρε βιώσιμες επενδύσεις... σε χαλεπούς οικονομικούς καιρού. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή βιομηχανική βάση προκειμένου να προσελκύουμε νέες επενδύσεις. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα, μια φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να έχουμε τι απαραίτητε βιομηχανικέ ικανότητε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των βιομηχανιών μα, ακολουθώντα συγκεκριμένε και γραμμέ όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, για παράδειγμα, προκειμένου να ενθαρρύνουμε περισσότερε επενδύσει. Μολονότι η έκθεση καλύπτει πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλούς τομείς, πιστεύω θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στις ε, επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν όσον αφορά τους ε, νέους. Η νεολαία στην Ευρώπη έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Έχουμε πάρα πολύ καλά μορφωμένους, καταρτισμένους νέους που αυτή τη στιγμή πλήττονται από την ανεργία, από την έλλειψη θέσεων απασχόλησης και είμαι σίγουρη ότι η συγγήτρια συμφωνεί με μένα καθότι προέρχεται από την Ελλάδα. Επομένως, οι τροπολογίες που θα υποβάλω θα έχουν σχέση με την απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να αυξήσουμε επίσης την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας όσον αφορά την ενέργεια. Πρέπει να επενδύσουμε επίσης σε πράσινες νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να προωθήσουμε και κάποιες αρχές φιλικές προς το περιβάλλον, θα πρέπει να συνοδεύουν τις πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν πιο βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες πράσινες, να πηγές ενέργειας και να εξαρτώμεθα λιγότερα από τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει επίσης πίσω από οποιαδήποτε στρατηγική να έχουμε συγκεκριμένες αρχές που θα καθοδηγούν την στρατηγική επενδύσεών μας και θα πρέπει να πετυχαίνουμε κάθε φορά μία γνήσια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα, το triple C, δηλαδή διασυνοριακή αποτελεσματικότητα φιλική προς το περιβάλλον και α, καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι επενδύσεις αυτές θα είναι τελικά και πιο αποτελεσματικές και πιο υποφελείς για όλους. Θα πρέπει οι επίσης να σέβονται το περιβάλλον, τα κοινωνικά κριτήρια, να δημιουργούν ε, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και θα πρέπει ουσιαστικά να είναι επενδύσει υψηλή ποιότητα. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανταγωνισμό φτηνών θέσεων εργασία. Θα πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα αξιοπρεπέ βιώσιμο οικονομικό σύστημα. Επομένω, όλε οι τροπολογίε μου θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν αυτή τη στιγμή το λόγο. Edward. Ο Βουλφ Κλίντ ε, θα παρουσίαζε ένα κείμενο, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Επομένως, μπορείς να μιλήσεις πρώτος. Um, Χαιρετίζω την έκθεση αυτή της κυρίας ε, Κράτσα Τσαγαροπούλου. Ε, μου φαίνεται πολύ ευχάριστη σε αυτή τη ε, στιγμή που μένεται ένας σκληρός οικονομικός χειμώνας έρχεται μια δροσιστική πνοή που μας κάνει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Βλέπουμε και από το παρελθόν ότι το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, προγραμματίστηκαν και άρχισαν να λειτουργούν ε, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαν την ε, προνοητικότητα να σκεφτούν ότι θα υπάρξει και μέλλον. Θα βγούμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα μπορέσουμε να κινηθούμε προς κάτι καλύτερο. Παρότι λοιπόν επικρατεί δρυμής χειμώνα, οι σπόροι κάτω από το χιόνι βλαστάνουν. Ας μην παρασυρθούμε λοιπόν από τις σκληρές συνθήκες του παρόντος χωρίς να σκεφτόμαστε το μέλλον. Πολύ καλό λοιπόν το ότι σκεφτόμαστε το μέλλον. Τώρα για το τι θα κάνουμε σε σχέση με κανονισμό κλπ. Ε, εμείς καλή την πίστη θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν τα προβλήματα του παρελθόντος. Βέβαια θα πρέπει να μην το παρακάνουμε για να μην ε, εμποδίσουμε την ε, πιθανή ανάπτυξη. Δηλαδή, όποιο ε, κανονισμό και αν εγκρίνουμε για την οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει ή που θα αφορά τη ρευστότητα ή που θα περιορίζει τις τράπεζες. Υπάρχουν πολλοί κανονισμοί στους οποίους αν το παρακάνουμε υπάρχει ο κίνδυνος να εμποδίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, την εξής κατάσταση. Η μία πλευρά ασχολείται με την εξυγίανση του προϋπολογισμού και τίποτα άλλο και η άλλη πλευρά μιλάει για ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Πού θα τη βρούμε όμως την ανάπτυξη αν δεν προκύψει από επενδύσεις. Άρα είναι σημαντικό όχι μόνο να μιλάμε για την ανάπτυξη, αλλά να μιλάμε και για αυτά που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, δηλαδή επενδύσεις. Και πρέπει να προετοιμάσουμε τις υποδομές, να προετοιμάσουμε το δυναμικό που θα προσελκύσει επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε πολύ σωστά. Είναι μια πολύ σημαντική και πολύ ισχυρή περιφέρεια με μεγάλο δυναμικό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε είτε μέσω της εσωτερικής αγοράς, είτε μέσω άλλου τομέα, με τους οργανισμούς ε, πιστοληπτικής ικανότητας, ε, με φορείς για την νεότητα, όλα θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα αυξήσει την ελκυστικότητά της για τις επενδύσεις, πράγμα το οποίο θα επιφέρει και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ δεν έχει έρθει και ο Σαμόζα. Εγώ εκ μέρους του ΟΑΛΤΕ λοιπόν ε, θα δώσω ένα σύντομο σημείωμα από τον σκιώδη συγητή τον Βολφ Κλίντς που χαιρετίζει ε, το σχέδιο έκθεση της κυρίας Κράτσα για την ε, ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Θεωρεί ότι η έκθεση θίγει πολλά πολύτιμα σημεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη που είναι σημαντικές προϋποθέσεις ούτως ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ελκυστική για επενδύσεις από από ε, έξω στο μέλλον. Ε, έχει και κάποιες συμπληρωματικές ιδέες από την πλευρά των φιλελευθέρων. Είναι ήδη πολύ ισορροπημένη η έκθεση αυτή, αλλά με κάποιες προσθήκες ε, κατά τη συνεργασία σας νομίζω το κείμενο θα μπορέσει να υποφεληθεί. Περιμένει λοιπόν και προσβλέπει τη συνεργασία μαζί σας και με τους σκιώδεις συζητητές στο μέλλον. Θα ήθελα και εγώ ίδια να κάνω κάποια σχόλια. Χαιρετίζω αυτή την προσέγγισή σας. Το βλέπετε σαν ένα βασικό οριζόντιο θέμα σε όλες τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για τη στρατηγική 2020. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει ε, να εξετάσουμε την ελκυστικότητα των επενδύσεων παράλληλα με όλο το νομοθετικό έργο που κάνουμε. Δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο ρυθμιστική νομοθεσία των αγορών, ούτε λέμε ότι δεν πρέπει να έχουμε ρυθμιστική νομοθεσία στην αγορά, αλλά πάντοτε πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι η επίπτωση αυτών που κάνουμε επί της ανάπτυξης, για να μην υπάρχουν ε, παρενέργειες και στην περίπτωση που υπάρχουν αθέλητες συνέπειες να ληφθεί κάποια εξισορροπιστική δράση. Και όπως λέει και ο Μισελ Μπαχνιέ, από πλευράς νομοθετικών προτάσεων η ομάδα του G20 έχει κάνει την προσπάθεια και τώρα πρέπει να περάσουμε στη φάση του να αναγνωρίσουμε τις επιπτώσεις επί της ανάπτυξης και να δούμε τι αθέλητες συνέπειες μπορεί να υπήρξαν ή να υπάρχουν και να τις αντιμετωπίσουμε. Να δώσουμε δηλαδή το μήνυμα ότι στην Ευρώπη είμαστε ανοιχτοί για επιχειρηματικό πνεύμα να μην δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι κατά των επενδύσεων. Ποιος θα ήθελε τον λόγο? Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κράτσα για την ε, εισήγησή της. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται βέβαια να προσέχουμε και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα παρόμοιο θέμα, γιατί η προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρώπη έχουν όλα αυτά να κάνουν με το κεντρικό θέμα της ανάπτυξης. Και πολλές φορές όταν μιλάμε για ανάπτυξη, έχουμε από τη μια μεριά ανάπτυξη και από την άλλη προβλήματα όσον αφορά τα και αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια είναι να καθίσει κάτω να συντάξει μια στρατηγική για την ανάπτυξη και να προσελκύσει επενδύσεις στην Ευρώπη. Και νομίζω κυρία Κράτσα ότι η έκθεσή σας πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά να πω ότι χρειάζεται να προσέξουμε δύο σημεία να δούμε το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας. Αναφέρθηκε η Ιρλανδία, παραδείγματο χάρη. Αλλά οι διάφορες χώρες, ε, εκτός από το δικό τους φορολογικό σύστημα, μπορούν να έχουν και διαφορετική πολιτική που προσελκύουν τις ξένες επενδύσεις και θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και η στρατηγική των επενδύσεων γίνεται μέσα από μια δουλειά που πρέπει να κάνει το ίδιο το κράτος πάνω σε πολλούς τομείς όπως στη δικαιοσύνη, στην παιδεία και θα πρέπει να αποφύγουμε και την υπερβολική γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε σε πολλά κράτη-μέλη. Όλα αυτά χρειάζεται να τα λάβουμε υπόψη μας στην έκθεση και η στρατηγική 2020 θα πρέπει να είναι κάτι το πιο συγκεκριμένο παρά ένα σκέτο κείμενο. Θα πρέπει να εφαρμοστεί όπως πρέπει η στρατηγική 2020 και οτιδήποτε έχει να κάνει με περισσότερη ανάπτυξη πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πάντως κρίνω θετικά την έκθεσή σας. Σβέν, βλέπω ότι έφτασες. Θέλεις να μιλήσεις, όχι. Υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Αν όχι, τότε δίνω το λόγο πάλι στην εισηγήτρια. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε και εσά προσωπικά και τους συναδέλφους για την παρέμβασή τους, για το, καταρχάς για το θετικό πνεύμα με το οποίο βρίσκουν, ε, βλέπουν αυτή την έκθεση, τόσο για τη σημασία της αυτή την πολιτική και οικονομική περίοδο, την κρίσιμη που διάγουμε στην Ευρώπη ε, και δεύτερον για τις επιμέρους παρατηρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι τονίστηκε ο ρόλος μας στο πλαίσιο το διεθνές. Αναφερθήκατε και εσείς στο G20 πώς η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει σε μια, στη διεθνή regulation και πώς πρέπει να δούμε αυτά τι επιπτώσεις έχουν στην ε, ε, οικονομική μας ζωή και την επενδυτική μας δραστηριότητα τις ε, ε, ε, ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια στρατηγική συγκεκριμένη και τις ευθύνες των κρατών μελών διότι πολλά πράγματα για το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, πιστεύω ότι και αυτό είναι το πνεύμα και της δικής μου έτσι, πρότασης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ε, τα, τα νέα καινοτόμα εργαλεία. Ε, έχω ήδη αναφερθεί στην έκθεσή μου στα, ευρωμόλογα έργων πως πρέπει να προωθήσουν ε, την επενδυτική μας δραστηριότητα. Άλλα πράγματα μπορούμε να εισάγουμε, τις επενδύσεις νέων για να τις να έλξουμε τους νέους. Έχω ήδη και εγώ κάποιες ιδέες. Ξέρετε, πολλές ιδέες δεν μπόρεσαν να χωρέσουν στο περιορισμένο πλαίσιο που έχουμε ως προς τις λέξεις και την έκταση. Έχω ε, το start-up, παραδείγματος χάρη, είναι μια ιδέα που θα την εισάγω με τροπολογία, πως πρέπει να αποτελέσει ένα αντικείμενο μελέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και το start-up κυρίως αφορά τους νέους και τα, καινοτόμα θέματα. Επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που τονίστηκε και που το, κάνει και το αναφέρει και η έκθεση ότι οι επενδύσεις είναι ένα οριζόντιο θέμα αλλά πρέπει να τύχουν και μια ιδιαίτερη συνεκτική προσέγγισης και επίσης αυτό που είπατε κυρία συνάδελφε για τη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης ε, είναι κάτι στο οποίο έχει υποχώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να το ανεχτούμε. Θα δώσει προστιθεμένη ευρωπαϊκή αξία σε πολλές περιοχές της Ένωσης. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά θα ενταχθούν εύκολα στο πλαίσιο που υπάρχει και είναι σημαντικό ότι όλοι συμφωνούμε για τη σημασία του θέματος και το πλαίσιο, στο πλαίσιο το οποίο παρουσιάζεται ήδη η πρότασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως είναι πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Η 26η Απριλίου το μεσημέρι είναι η ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών. Στις 30 Μαΐου θα εξετάσουμε αυτές τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 31 Μαΐου στην Επιτροπή και η έκθεση θα πάει στην Ολομέλεια στην πρώτη σύνοδο του Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε όλους που συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Ο εισηγητής μας για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει δεν είναι διαθέσιμος μέχρι τις 11.30. Έτσι προβλεπόταν ε, τουλάχιστον στη μερίσια διάταξη να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το CRD4. Έχουμε λοιπόν 45 λεπτά στην διάθεσή μας, μπορούμε να διακόψουμε και όσοι συμμετέχετε στη συζήτηση για το CRD4 επιστρέψτε παρακαλώ πολύ λίγο πριν τις 11.30. Κάνουμε λοιπόν διάλειμμα μέχρι τις 11.30. Ευχαριστώ. από πολλά και φορά. Ευχαριστώ.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

αυτό και δεν υπάρχει που να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

και να φτάσουμε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

AUTHORWAVE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 Σας ευχαριστώ.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 Right, welcome, welcome back Ας συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Όσοι είναι να συμμετάσχετε, μπείτε σε παρακαλώ πολύ στην αίθουσα. Περνάμε τώρα στη συζήτηση για το CRD4, Οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσει, δεύτερη ενταλλαγή απόψεων για τις ε, τροπολογίες ο εισηγητής και οι σκιώδεις ε, εισηγητές θα μπορέσουν να συζητήσουν το πώς προχωρούν τα πράγματα όσον αφορά την εξέβρεση συμβαστικών τροπολογιών. Νομίζω ότι σε αυτό θα εστιάσουμε. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Ότμαρ για να μας πει κάποια αγωγικά πράγματα, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να σας παρουσιάσω τις γενικές τάσεις. Δεν είναι μια γενική συζήτηση για την ΟΚΑ 4 και τη Βασιλεία 3. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση των συζητήσεων με τους σκιώδεις εισηγητές και τι εξελίξεις υπάρχουν τι πιθανές συμβιβαστικές τροπολογίες υπάρχουν. Επ' αυτόν θα ήθελα να σας ενημερώσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Γιούλια Κρέτ, συνεργάτειά μου, και τους συνεργάτες ε, της Γραμματείας και τους κοιόδης εισηγητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για την ε, πληρέστατη συνεργασία που είχαμε στις δραστηριότητες της Επιτροπής. Χωρίς την τεχνική συνεργασία όλων των συνεργατών δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και τις χρονικές δυσκολίες και τις δυσκολίες περιεχομένου αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πραγματικά λοιπόν ειλικρινά. Κάτι ακόμη τώρα για την Επιτροπή μας οι Υπουργοί Οικονομικών έχουν άρει αυτά τα θέματα σε ομάδες εργασίας στο δικό τους επίπεδο. Αναμένουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου και χαιρόμαστε ότι, διότι υπάρχει 3 Μαΐου μια ειδική συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών, διότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, χρειαζόμαστε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο ε, κοινή θέση με την επαρκή βάση για να μπορέσουμε να έχουμε διαπραγματευτικές θέσεις. Ανεξάρτητα από τα χρονοδιαγράμματα και τις δυσκολίες του Συμβουλίου, εμείς θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και τις γραμμές μας και τον ε, Ιούνιο, το αργότερο τον Ιούλιο θέλουμε να μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια. Έχουμε κάνει πολλές ε, συζητήσεις ε, μεταξύ σκιωδών εισηγητών και χτες στη συνάντηση σκιωδών εισηγητών συμφωνήσαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε κάθε μέρα συζητήσεις σε επίπεδο συνεργατών και στο τέλος της εβδομάδος στο Στρασβούργο θα κάνουμε το επόμενο την επόμενη πολιτική συζήτηση μεταξύ σκιωδών εισηγητών και θα αξιολογήσουμε τις εξελίξεις. Δουλεύουμε συνεχώς με τους σκιώδεις και με τους συνεργάτες μας και με όλους ε, τους ε, συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες ούτω ώστε να μπορέσουμε κεφάλαιο προς κεφάλαιο και κάθε συμβιβαστική λύση να τα διαπραγματευτούμε και προσπαθούμε να κρατήσουμε το ε, εύρος το οποίο θέλουμε να έχουμε σε μια έκθεση πρωτοβουλίας για να μπορεί να γίνει η συζήτηση αυτή στο σωστό πεδίο. Σήμερα θα ήθελα να σας αναφέρω πέντε δύσκολα σημεία στα οποία προσπαθούμε να έχουμε μια συμβιβαστική λύση. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις πρόοδους που έχουμε επιτύχει. Πρώτον, όσον αφορά τη στάθμιση κινδύνου. Νομίζω ότι εκτός από πολύ μικρές λεπτομέρειες κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η χορήγηση πιστώσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνεται μέσω της ε, πρότασης της Βασιλείας η διευκόλυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασίζεται σε δύο στοιχεία στην πιθανή συμβαστική λύση. Πρώτον, μία μείωση, μείωση ε, τη στάθμιση κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που ονομάζουμε balancing factor, είναι μια μείωση από το 75% στο 50%. Μείωση λοιπόν κατά το 1 τρίτο για τις ε, πιστώσεις που χορηγούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερο στοιχείο για τη μείωση του κινδύνου είναι η αύξηση των κατοφλίων. Το έχουμε ζητήσει στην έκθεση όπως γνωρίζετε και έχει ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξέταση των δυνατοτήτων που υπάρχουν μέχρι το Σεπτέμβριο θα υποβάλουν κάποια έκθεση. Εμείς θέλαμε την πρόταση μέχρι το Μάιο και αν δεν έχουμε την πρόταση μέχρι το Μάιο, θα ανοίξουμε την πόρτα στη διαπραγματευτική διαδικασία μέσω του Κοινοβουλίου για να έχουμε διπλασιασμό του κατοφλίου από 1 εκατομμύριο στα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι βέβαια η τελευταία λέξη, γιατί θα πρέπει ε, να εξετάσουμε όλα τα σχετικά στοιχεία, μήπως τυχόν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη αύξηση. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο σημείο για την αύξηση του κατοφλίου από το 1 εκατομμύριο στα 2 εκατομμύρια. Και αν υπάρχει δυνατότητα θα αυξήσουμε το κατόφλι ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το πρώτο σημείο αφορούσε το, τη στάθμιση κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με, αυτά τα δύο, με αυτούς τους δύο πυλώνες που ανέφερα. Δεύτερο κεφάλαιο, ρευστότητα. την ε, περίοδο αξιολόγησης θέλουμε να την ε, θέσουμε κατά τρόπο να είναι αποτελεσματική και θέλουμε να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία προτείνονται στις τροπολογίες των συναδέλφων. Θέλουμε να έχουμε πράξεις κατεξουσιοδότηση για το LCA. περίοδος αξιολόγησης των ρευστών θα πρέπει να μπει ε, κατά τρόπο να είναι αποτελεσματική με βάση αυτά τα οποία προτείνουν οι συνάδελφοι στις τροπολογίες και πράξη κατεξουσιοδότηση. Τρίτο κεφάλαιο το οποίο εξετάζουμε όσον αφορά τις συμβαστικές προτάσεις ρυθμίσεις ε, για τις ε, απολαβές. Αυτό είναι ένα στρατηγικό ζήτημα. Θέλουμε να δούμε πώς, θα πάνε οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό όριο και συζητάμε το κατά πόσο θα καθιερώσουμε ένα απόλυτο ανώτατο όριο στους πιο υψηλούς μισθούς. Στη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό το θέμα. Θέλουμε μια πολύ αυστηρή ρύθμιση. για να έχουμε μια μεταβλητή ένα προς ένα. Τέταρτο κεφάλαιο Έχουμε ένα ε, συμπληρωματικό αποθεματικό στη Βασιλεία για το συστημικό κίνδυνο. Και το πρόσθετο απόθεμα μπορεί να είναι από 1 έως 5% φτάνοντας μέχρι 10%. Τελευταίος τομέας, τελευταίο κεφάλαιο για τις τροπολογίες είναι η τροποποίηση των ρυθμιστικών διατάξεων ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο. και στις προσεχείς εβδομάδες θα, προσκαλέσουμε και τον πρώην Επίτροπο πολύ Κάνεν που είχε μια ομάδα εργασίας για τις τραπεζικές διαρθρώσεις για να δούμε τι καλύπτεται στη Βασιλεία σε σχέση με τις τραπεζικές διαρθρώσεις. Ανεξάρτητα από αυτό, προσπαθούμε να δούμε τι διαφοροποίησεις μπορούμε να έχουμε μέσα στη Βασιλεία χωρίς ε, να δημιουργείται κανένας κίνδυνος. Στόχος μου παραμένει, και δεν ξέρω αν αυτό αρέσει σε όλους, θέλουμε να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τράπεζες που θα ισχύει για όλους. Θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα, αλλά θα ισχύει για όλους. Και θέλουμε να διαμορφώσουμε μια εσωτερική αγορά, να σταθεροποιήσουμε την χρηματοπιστωτική αγορά, δημιουργώντας βέβαια κάποια ευελιξία, αλλά αυτό που θέλουμε είναι μια σωστή χρηματοπιστωτική αγορά. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα θεσπίσει. Δεν θέλουμε να τεθεί σε κίνδυνο το single roll book. Όσον αφορά το συντελεστή μόχλευσης και το NSFA, είναι δύο τομείς όπου πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαφοροποίηση και θα υποβάλουμε προτάσεις και θα δούμε αν υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους να είναι δυνατή μια τέτοια διαφοροποίηση λαμβάνοντας υπόψη και τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι. Τώρα από εδώ και πέρα σας είπα ότι για την επόμενη εβδομάδα κάθε μέρα θα γίνονται τεχνικές συζητήσεις και την Παρασκευή θα γίνει η επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, λαμβάνοντας υπόψη όσα θα, έχουμε, θα έχουν συζητηθεί στις τεχνικές συναντήσεις. Και έχουμε υποσχεθεί ότι μέχρι την Τετάρτη ή την Τετάρτη θα γίνουν οι συζητήσεις ούτως ώστε να καλύψουμε τις επιθυμίες ε, όλων και να συμφωνήσουμε μεταξύ όλων των σκιωδών εισηγητών τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το οποίο δεν κάνουμε είναι συζητήσεις με λόμπι και με ομάδες συμφερόντων, γιατί θέλουμε να επικεντρωθούμε στη δουλειά που έχουμε με τις 1500 τροπολογίες για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή βάση για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Και όταν θα έχουμε κοινή θέση, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ούντο Μπούλμαν μπορεί να μας μιλήσει εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Κάρας που είναι ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ γιατί έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και ευχαριστώ και για την έκθεση που μας παρουσίασε σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο σε αυτή την ομάδα εργασίας των σχεδόν εισηγητών για αυτό το νομοθετικό κείμενο είναι και αυτό μπορώ να το πω εγώ που έχω συνεργαστεί είναι ότι υπάρχει καλή βούληση. Και επειδή υπάρχει κοινή θέληση, ενθαρρυνόμαστε όλοι να προχωρήσουμε. Πιστεύουμε όλοι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία και να συνεισφέρουμε με θετικό τρόπο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεως. Και θέλω να τονίσω τα σημεία τα οποία θεωρούμε σημαντικά και αυτά τα οποία εμείς ως ομάδα των σοσιαλδημοκρατών έχουμε προτείνει σε όλους τους συναδέλφους και στον εισηγητή τον Ότμαρ Θέλω να αναφέρω κάποια σημεία που για τη δική μας πολιτική ομάδα είναι περισσότερο σημαντικά. δεν έχουμε εξαιρέσεις μέχρι τώρα, δηλαδή ο τραπεζικός τομέας δεν μπορεί να καλύψει τις δικές του ελλείψεις και να τα φορτώσει στους ώμους των φορολογου... στις πλάτες των φορολογουμένων. Δεν θέλουμε πια να χρηματοδοτούμε την κακή διαχείριση. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για μας γίνεται μια πολύ ζωντανή συζήτηση και το ανέφερε και ο Ότμαρ Κάρας για το πώς μπορούμε να έχουμε ακριβή διαφοροποίηση για τους φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος που είναι αυτοί που προκαλούν κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτή τη διαφοροποίηση πρέπει να την κάνουμε δεν έχουμε βρει ποιο είναι το κατάλληλο μέσο για να το κάνουμε. Έχουμε πει ότι μπορεί να είναι το ύψος του ισολογισμού. Άλλοι λένε ότι πρέπει να ταξινομήσουμε τις τράπεζες ε, σε διάφορες κατηγορίες. Έχει κάποιες προτάσεις ο εισηγητής επί του θέματος. Τελικά θέλουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή μέθοδο διαφοροποίησης. Συνεχίζεται η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε ε, να καταλήξουμε σε μια λύση. Αν θα είναι οι απαιτήσει κεφαλαίου, αν θα είναι ε, ε, οι απαιτήσει ρευστότητας, θα δούμε ποια θα είναι η μέθοδος. Πάντως, όλοι επιθυμούμε να έχουμε καλύτερη διαφοροποίηση, να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν τον κίνδυνο και τι σημαίνει υπεύθυνη άσκηση τραπεζικής λειτουργίας, κάτι το οποίο να είναι πολιτική και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε πού βρίσκονται αυτοί που προκαλούν τους μεγάλους κινδύνους, ώστε να μην μπορεί κανείς να κρυφτεί πια. Έχει δίκιο ο Ότμαρ Κάρας που λέει ότι δεν δημιουργούμε νέα τραπεζική δομή μέσω αυτής της οδηγίας. Δεν δημιουργούμε, αλλά μπορούμε να προετοιμάσουμε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πορεία προς την οποία έχουμε ξεκινήσει. Δεύτερο σημείο. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό ε, ισχύει για κάποια σημεία ε, ε, που ε, παραμένουν σε κρεμότητα, που είναι ακόμη ανοιχτά από την ε, ΟΚΑ 3, ο εισηγητής είναι πρόθυμος να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ θα έχουμε μια διένεξη με το Συμβούλιο. Αυτό νομίζω διαφαίνεται ήδη. Στο θέμα αυτό το Συμβούλιο δεν μπορεί να δράσει, δεν μπορεί να τηρήσει το, το χρονοδιάγραμμά του αλλά φαίνεται ότι τα καυτά θέματα που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο να τα αντιμετωπίσει, όπως είναι οι απολαβές και ο τρόπος διαμόρφωσης των απολαβών και των αποδοχών. Χαίρομαι που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με το Συμβούλιο και το περιμένω πώς και πώς, γιατί νομίζω ότι και τα μέσα ενημέρωσης και οι εκλογείς θα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το θέμα, να δουν ποιος βρίσκεται σε ποια πλευρά και ποιος τελικά αναλαμβάνει την ευθύνη ή ποιος παρεμποδίζει τις προτάσεις που υποβάλλονται. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο το Κοινοβούλιο θα έχει πολλά να πει. Ένα βασικό σημείο εδώ σε αυτόν τον κανονισμό είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληρώνουν τα σφάλματα. Μπορούν να γίνουν πολλά σε αυτό τον τομέα. Ανέφερε ο Ότμαρ Κάρες κάποιες προτάσεις και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή στην πράξη να δούμε πώς μπορούμε ε, να ε, έχουμε μέτρα περισσότερο φιλικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δική μας πολιτική ομάδα έχει προτάσεις και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια κοινή συμβαστική λύση. Τέλος, ένα από τα μεγάλα θέματα, αν θα έχουμε μέγιστη ή ελάχιστη εναρμόνιση. Ο εισηγητής ε, λέει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορούμε να είμαστε αρκετά ευέλικτοι για να ε, επιτρέψουμε στις διάφορες χώρες να τηρήσουν τη γραμμή που θέλουν να, τηρήσουν. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τη σωστή συμβιβαστική τροπολογία τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας πω ποιοι είναι οι ομιλητές. Έχουμε μισή ώρα μπροστά μας. Εγώ ίδια, Φίλιπ Λάμπερτ από τους Πρασίνους, Jean Paul Gauzès. Βλέπω και την Ελίσσα. Να σας ε, υπενθυμίσω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν θα πρέπει να καλύψουμε αυτή τη στιγμή όλες αυτές τις χιλιάδες των τροπολογιών. Θα κάνουμε πάντως ό,τι μπορούμε στο διαθέσιμο χρόνο που έχουμε. Ναι, ναι, θα μιλήσετε, μην ανησυχείτε. Εκτός μικροφώνη παρατήρηση της κυρίας Μπερές. Ακούσατε πάντως τι σας είπε ο εισηγητής. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, θα ήθελα και εγώ να πω κάποια πράγματα όσον αφορά την εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταρχάς, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τις προτάσεις που έχουν γίνει για την ε, εξισορρόπηση του κινδύνου, για τη στάθμιση του κινδύνου, Έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες, οι οποίες βρίσκουμε ικανοποιητικέ, δημιουργούν έναν συμπληρωματικό μηχανισμό, όπου φαίνεται τελικά ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο κεφαλαίων, αν δεν λειτουργήσει το σύστημα το οποίο προβλέπεται. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα, λοιπόν, ένα συμπληρωματικό ε, μηχανισμό, στον οποίο μπορούμε να καταφύγουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του 443α, αυτού του άρθρου δηλαδή, όπου έχουμε και όλα τα ε, εργαλεία της ε, μακροπροληπτικής εποπτείας. Δεν απαραίτητο ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, για τις προτάσεις που γίνονται για τη ρευστότητα τώρα. Συμφωνώ εν γέννη με τις ε, σχετικές προτάσεις θα έλεγα όμω ότι υπάρχουν και κάποιε άλλε τροπολογίε που δεν έχουν ακόμα εξεταστεί. Για παράδειγμα, η δική μου τροπολογία, υπαριθμών 97, όπου λέω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για ένα επιπλέον διαθέσιμο κεφάλαιο το οποίο θα μπορεί να υπάρχει. Όσον αφορά τώρα τις κατεξοδότηση πράξης για να εισαχθούν αυτές οι προτάσεις, Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ τις πιθανές ε, μεθοδολογίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Να δούμε πώς να αναπτυχθούν οι μεθοδολογίες αυτές και πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα στη μόχλευση και το NSFR. Οι προτάσεις αυτές βρίσκονται αυτή τη στιγμή μόνο σε ρήτρες αναθεώρησης και αν προχωρήσουμε μέσα σε ένα χρόνο με κατεξοδότηση πράξη, θα ήταν καλύτερο ορισμένες από τις ρήτερες αυτές να περάσουν στο άρθρο 402, αντί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 481. Επίσης, ενδεχομένως να έρθουμε σε αντιπαράθεση με μια άλλη νομοθετική πράξη, όταν χρησιμοποιούμε τις κατεξοδότηση πράξεις. Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια ότι θα πρέπει να, μάλλον, όταν, άμα να χρησιμοποιήσουμε κατεξότηση πράξη, πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αν δεν υπάρχει κάποια πρώτερη νομοθεσία. Αν προκύψει λοιπόν μια πλήρης νομοθεσία νωρίτερα, τότε θα καλυφθούν τα πράγματα μέσω της νομοθεσίας αυτής, διαφορετικά θα πρέπει να καταλήξουμε στις κατεξοδοτήσεις πράξεις. Θα ήταν πολύ περίεργο να έχουμε ένα πλήρε νομοθετικό πακέτο και να έπρεπε να δεσμευτούμε παράλληλα από τι κατεστωτέ πράξει. Τώρα, για το άρθρο 404. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να επιφέρουμε κάποιες ε, τροποποιήσεις. Δεν νομίζω ότι οι ορισμοί που παρέχονται εδώ πέρα όσον αφορά το eligible collateral σε σχέση με τις κεντρικές τράπεζες έχουν αντιμετωπιστεί σωστά. Γι' αυτό το λόγο έχω αποβάλει μια σχετική πρόταση μέσω, της, μέσω μιας τροπολογίας μου. Επίσης, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να έχουμε όλα αυτά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 404 σημείο 3. Είναι απαραίτητο να τηρήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να πούμε ή το ένα ή το άλλο. Και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένους ορισμούς όσον αφορά την έννοια του Repurchased Agreement. για τις συμφωνίες επαναγοράς, για τα ρέπος. Και όσον αφορά τώρα το σημείο 5, ξέρω ότι εδώ πέρα θέλετε να λάβετε υπόψη σας την τροπολογία 106.1 του Φίλιπ Λάμπερτ. Νομίζω πάντως ότι δεν θα ήταν απαραίτητο να περιοριστούμε εδώ πέρα σε συγκεκριμένα ποσά 250 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα. Αν έχουμε τις απαραίτητες ρήτρες αναλογικότητας που άλλωστε προσπίζονται από το, από το 1061, από τροπολογία 1061, τότε αυτό μας καλύπτει. Και θα προτιμούσαμε να παραμείνει μέσω τροπολογίας η αλλαγή αυτή. Να πω κάποια πράγματα όσον αφορά το μέγιστο ή κατώτατο ποσό. Εργαζόμαστε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα εργαλεία αυτά της μακροπροληπτικής εποπτείας θεωρώ ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο μέσο προκειμένου να καταφέρουμε να προσαρμόζουμε τις σταθμίσεις κινδύνου στα πλαίσια ενός κράτους μέλους, ιδίως για ζητήματα όπως το residential property, όπως δηλαδή τα κεφάλαια τα οποία σχετίζονται με τα κίνητα που πολλές φορές οδηγούν σε φούσκες. Και σε ευρωπαϊκό όμως επίπεδο θα πρέπει να ισχύουν κάποιες συνθήκες ex post και ex ante. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν παράλληλο μηχανισμό και αν αυτό μπορεί να γίνει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένω μέσα σε τρει μήνε να σα πούνε ότι δεν θα πρέπει να καταλήξετε σε ένα τέτοιο μηχανισμό. Νομίζω πάντως, τουλάχιστον στη δική μου την ομάδα, ότι είμαστε γενικά απογοητευμένοι, είτε είμαστε υπέρ του ενός επίπεδου, του κατώτατου, είτε υπέρ του ανώτατου επίπεδου. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια κάποια μέση λύση. Αυτά είχα να πω. Όσον αφορά τις τροπολογίες που κατέθεσε η δική μου πολιτική ομάδα, μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον Φιλίπ. Ευχαριστώ, Σάρων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νότμαρ. Όλοι ευχαριστούν τον Ότμαρ, αλλά πραγματικά εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτό το δύσκολο ε, έργο ο Ότμαρ. Εκτιμώ ιδιαίτερα και τον ανοιχτό του χαρακτήρα και την προθυμία για συμβαστικέ λύσει. Λοιπόν, τρία σημεία. Πρώτον, διαφοροποίηση. Στι τροπολογίε μα λέμε ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών σε τρει κατηγορίε. Σύφη, ε, Ε, ουσιαστικές τράπεζες και όλα τα άλλα τα ενδιάμεσα. Υπάρχουν κριτήρια που μας επιτρέπουν να πρέπει να υπάρχουν κριτήρια που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε τη διαφοροποίηση και πρέπει από τις κατηγορίες αυτές να προκύπτουν απαιτήσει όχι μόνο για τη μόχλευση και τη ρευστότητα αλλά και για το κεφάλαιο και πρέπει να είναι διαφοροποιημένα τα κριτήρια γιατί υπάρχουν διαφορετικά προφίλ κινδύνου. δεν είναι μόνο ΣΥΦΙΣ, ε, αλλά όλες ε, οι τράπεζες γενικότερα αυτές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό πιστεύω εγώ. Συνεχίζεται όμως η συζήτηση. Σχετικά με τη ρευστότητα, θα ε, έχουμε πράξεις κατά για το LCR και για το NSFR, συμφωνώ με τη Σάρων. Θέλουμε να έχουμε και περιορισμούς για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κινητών αξιών και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύει κατά τον ίδιο τρόπο για το δίκτυο ρευστότητα των ΟΣΕΚΑ. Ακόμη επιμένουμε για την τροπολογία 1015 για την ε, κάλυψη κινδύνου και το κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας. Όσον αφορά τον κίνδυνο δημοσιοποίησης, επιμένουμε. Πιστεύουμε ότι η δημοσιοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο κλάδος ήδη εφαρμόζει το 90% του NSFR. Δεν είναι λοιπόν πολύ μακριά. Τους δίνουμε τη δυνατότητα, τη χρονική δυνατότητα να φτάσουν το 100%. Άρα ας επιμείνουμε γιατί ξέρουμε ότι ο κλάδος ήδη κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σχετικά με τον δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της διαφοροποίησης θα θέλαμε να το επιτύχουμε. Θα το προτιμούσαμε από το να παίζουμε με το δίκτυ ε, κινδύνου. Ο πραγματικός κίνδυνος για το δανεισμό των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να είναι 50 ή 75% ή οτιδήποτε πούμε, αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, πραγματικά στοιχεία και όχι απλώς το ότι θέλουμε να ευνοήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποια φούσκα. Τώρα, για γιατί ε, θέλουμε να δούμε μία ρήτρα για την αξιολόγηση κινδύνου, για το πώς αξιολογεί ο κίνδυνος από τους διάφορους φορείς της αγοράς. Ο σκοπός μας είναι κάποια πειθαρχία στην αγορά. Ακόμη θα θέλαμε οι απαιτήσει κεφαλαίου να σχετίζονται με τους κανόνες που ορίσαμε. Θέλουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να είμαστε κάτω από τα πρότυπα του, της Βασιλείας 3. Λέμε ότι θα πρέπει οι κατουσίαν τράπεζες να είναι στο Βασιλείας 3 και η ΣΥΦΙ θα πρέπει να είναι στο πιο πάνω όριο. Δεν λέμε ότι πρέπει να έχουμε λιγότερη πειθαρχία, αλλά θα πρέπει ε, να τη χειριστούμε κατά τον πιο ευνοϊκό τρόπο. Για τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να μας δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης όχι στη μέση της κρίσης αλλά στο δυνατόν νωρίτερα. Και για τα αποθέματα πρέπει να δούμε για τι ε, ε, αναλογία μιλάμε όταν μιλάμε για ε, αναλογία του ΑΕΠ και θα πρέπει να έχουμε μια σταδιακή προσέγγιση για το κατόφλι που θα ενεργοποιεί το απόθεμα. Νομίζω ότι στον κλάδο κάτι πρέπει να γίνει και για την πολιτική αποδοχών. Έχουμε προτείνει και εμείς κάτι και οι σοσιαλιστές έχουν προτείνει κάτι. Ένα προ 40 ή κάτι τέτοιο νομίζω θα ήταν το λογικό. Ένα θέμα που ακόμη δεν έχουμε θίξει είναι το shadow banking. Θέλουμε να είναι περιορισμένη αυτή η δραστηριότητα και να υπάρχει ένα ανώτατο όριο στην νομοθεσία και ελπίζω ότι κάτι τέτοιο θα μας θα το βρούμε μπροστά μας στις συζητήσεις που κάνουμε για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, πολύ, Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σύντομος θα είμαι. Είναι ανοιχτή συζήτηση και δεν θα πρέπει να δούμε τώρα άλλες λεπτομέρειες, αλλά να συγχαρώ για όλη την εργασία αυτή τη δουλειά. Έχει πολύ ακόμα μπροστά του και τον υποστηρίζω στα διάφορα σημεία τα οποία αναφέρθηκε, αλλά αντιμετωπίζω κάποιο προβληματάκι σχετικά με τις κατεξοδότηση πράξεις. Στο IFMD αυτά που έχω δει, τι μου δείχνουν, ότι η συζήτηση για τις κατεξοδότηση πράξεις επιτρέπουν σε μερικούς να ξαναξεκινήσουν μια συζήτηση για το αρχικό κείμενο και μάλιστα προς τις δύο κατευθύνσεις. Όσοι είναι στις ομάδες πίεσης λένε «Α, προδίδεται το αρχικό κείμενο με επιπλέον απαιτήσει και ταυτόχρονα τι προσπαθούν να κάνουν, να ελαφρύνουν τα κατάσταση και τα πράγματα». Κάπως μπερδεμένο είμαι τώρα σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, με αυτά τα στοιχεία. Από τη στιγμή που πρόκειται για το LCR, ίσως θα πρέπει κανείς να το ρωτηθεί μήπως χρειάζεται και εδώ να έχουμε μια συναπόφαση πριν να ρυθμιστούν οριστικά τα πράγματα. Πρέπει να το σκεφτούμε και με την σημερινή πείρα που διαθέτουμε για τις κατεξοδότηση πράξεις, εντάξει, και τώρα για το IFD, η ΤΑΔΕ, άλλη εφημερίδα λένε ότι σκοτώνουμε τα οικονομικά αυτά θέματα και θα πρέπει οι σκεδοσηγητές να το αναρωτηθούν και για τις αμοιβέ. Εντάξει, συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητού. Ε, είναι μεταθάνατο νίκη, πύριος νίκη, γιατί ε, για τη Βασιλεία Τρία. Είχα πει τότε στον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών ότι αυτή η εγγραφή αυτής της συμφωνίας δεν ήταν ε, ε, καλύδα, είπαν ναι, ένα fair play και βλέπουμε ότι όταν γίνονται τα πράγματα κλείνουν ακόμα περισσότερο οι πόρτες και αποτελεί ένα πολύ καλό μάθημα αυτό που συνέβη. Ευχαριστούμε πολύ, Κάρι. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ και εγώ ιδιαίτερα το πολύ δύσκολο αυτό καθήκον το οποίο είχε αναλάβει ο Ότμαρ Προσπαθεί να διατηρήσει την σωστή ταχύτητα στην επεξεργασία του κειμένου, αλλά είναι και πολύ αυστηρό με το περιεχόμενο. Αν δούμε πώ εξελίσσονται τα πράγματα στο Συμβούλιο έχουμε την εντύπωση ότι θα καταλήξουμε σε ένα κοκτέιλ, σε ένα μείγμα εθνικών τελικά συμφερόντων. Επομένως, είναι δική μας υποχρέωση να ακολουθήσουμε με ένα λογικό τρόπο την ευρωπαϊκή προσέγγιση, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε και μια σωστή ταχύτητα. Και νομίζω ότι εδώ πέρα τα όσα λέγονται για το ECRB, οι κατευθυντήριες γραμμές δηλαδή για τα αποθέματα ασφαλείας, είναι, ε, οι σχετικές προτάσεις είναι πολύ καλές. Επίσης όμως και σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, καθώ επίση και με τα όσα γίνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική διαπραγματευτική στάση απέναντι στο Συμβούλιο, όσον αφορά το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν τόσο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Να αναφερθώ σε τρία επιμέρου ζητήματα. Πρώτον, LCR, αναλογία κάλυψη ρευστότητα. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε ρήτρε μέσα στην νομοθεσία την οποία θα εγκρίνουμε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία πράξη, αν θα πρέπει να έχουμε μία συνομοθεσία εδώ πέρα, θα πρέπει να έχουμε ε, κατεξοδότηση πράξης. Θα πρέπει πάντως να λάβουμε υπόψη μας και τα όσα προβλέπονται για τις εξασφαλίσεις υψηλής ποιότητος. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα κριτήρια ποιότητος όσον αφορά το haircut, το κούρεμα, καθώς επίσης και συγκεκριμένες προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε αξιόγραφα τα οποία να είναι υψηλής ποιότητος και αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσα από την αναθεώρηση. Συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά τι αποδοχές. Συμφωνώ επίσης και με τη διαφοροποίηση που πρέπει να γίνει όσον αφορά διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην αναθεώρηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας της, τη δανειοδότηση που προέρχεται από τις δημόσιες τράπεζες και το δημόσιο τομέα. Όσον αφορά τώρα τα ΣΥΦΙΣ, πρέπει να δούμε εδώ πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές κατηγορίες Κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω, ενδεχομένω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Για ποιο λόγο θα πρέπει να δώσουμε διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη για να επιβάλλουν ένα επιπλέον 10% όσον αφορά το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου. Μπορείτε να μου το απαντήσετε ενδεχομένω αυτό το ερώτημα αργότερα. Πίτερ Ζήμον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάρας, για την παρουσίαση των γενικών γραμμών συμβιβαστικών λύσεων όπω διαγράφονται. Έχω δύο ερωτήσει. Πρώτον, για τη στάθμιση κινδύνου για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, Είπατε ποια θα είναι η γενική κατεύθυνση. Μιλήσατε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η Επιτροπή στην στάθμιση κινδύνου μίλησε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τα φυσικά πρόσωπα. Ε, Κάποιο λόγο θα υπάρχει αυτό. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τουλάχιστον ε, στο βαθμό που ασκούν τη δραστηριότητά του ω φυσικά πρόσωπα. Βλέπω πόσε επιχειρήσεις υπάρχουν στη χώρα μου τουλάχιστον μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι επιχειρήσεις φυσικών προσώπων και δεν έχουν καθόλου τον ίδιο κίνδυνο όπως ε, οι ανώνυμες εταιρείε ή η ΕΠΕ. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να ληφθούν υπόψη και τα φυσικά πρόσωπα και η στάθμιση κινδύνου σε αυτές τις ε, περιπτώσει. Να μην επιβαρύνονται ε, από κίνδυνο. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο δεν αναφερθήκατε. Και για τις περαιτέρω συζητήσεις μας ε, θα ήθελα να λάβουμε υπόψη μας ε, για ε, τις στεγαστικές εταιρείες και η Επιτροπή ε, έχει λάβει υπόψη σε αυτό το θέμα και σκέφτεται μια σχετική αύξηση. Είναι ιδιαίτερα ε, κειμενόμενη η αγορά των ακινήτων αυτή τη στιγμή και ε, έχω υποβάλει τροπολογίες και μεγάλη μου χαρά θα τα συζητήσουμε στις περαιτέρω συζητήσεις μας για τις συμβαστικές τροπολογίες. Θέλουμε να έχουμε κάτι το σταθερό για τα επόμενα χρόνια για να τη δυνατότητα και σε κάποια μείωση της, αγοράς, της στεγαστικής αγοράς. Αυτό έχει και ένα φορολογικό υπόβαθρο. Ε, υπάρχει φορολογική επίδραση στις ε, αγορές με μεγάλη αύξηση του τομέα των ακινήτων. Όταν θα υπάρχει λιγότερη θα υπάρχουν λιγότερες, ε, λιγότερη κεφαλή, μικρότερη κεφαλιακή επάρκεια ε, για την ε, αγορά κινήτων, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα η αγορά κινήτων, η στεγαστική αγορά, να κινηθεί προς μια πιο σταθερή κατάσταση. Υπερβάνος έχει το λόγο. Αγαπητοί Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζω τις γνώσεις ε, του κύριου Καράς, ε, αλλά χάνει όταν έχουμε πάνω από χίλιες τροπολογίες ε, κάπως. Και θα ήθελα να τον βοηθήσω να του προτείνω χρήσιμα πράγματα της διαπραγματεύσης. Δεν ξέρω τις συμβαστικής τροπολογίες ούτε και η μεσκιώδη συγγήτρια. Πέρα από τα πέντε συμβαστικά που είπε ο συγγητής... Νομίζω ότι σιγά σιγά κατά την επεξεργασία της τοποθέτησης του Κοινοβουλίου θα έχουμε δυνατότητα να επανέλθουμε και σε άλλα σημεία που δεν υπησέρχονται σε αυτά τα πέντε που συμφωνήθηκαν και τότε θα ήθελα τότε να παρέμβω και να τονίσω μερικά πράγματα που θεωρώ σημαντικά και που θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός μιας πρώτης δέσμης ε, από ισχυρές προτάσεις του Κοινοβουλίου. Ο Φιλίπ Λαμπέρ είπε για το Shadow Banking System και νομίζω ότι υπάρχει και ο μηχανισμός ανταγωνισμού σχετικά με τη Βασιλεία. Τι γίνεται, αν βάζουμε το πράγματα έτσι, θα πρέπει να το δούμε και το shadow banking system, αλλά και πώς θα εφαρμόζεται η συμφωνία της Βασιλείας στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και όπως και Ορισμένοι από εμά κοιτάζουν προ τα εκεί, πέρα από τον Ατλαντικό. Θα πρέπει πάντω σίγουρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο να τοποθετηθούμε. Δεύτερος γεμικός προσανατολισμό τώρα. Πώς θα κατανεμηθούν όσο γίνεται καλύτερα τα κεφάλαια λάθος θα ήταν ε, να περάσουν αυτά τα μέτρα της Βασιλείας χωρίς να διορθώσουμε ε, προς τα που στοχεύουμε σχετικά με τη χρήση των χρημάτων. Πες δεν είναι ατέλειωτα τα χρήματα που έχουμε στην Ευρώπη. Γιατί μόνο είναι αποτελεσματική Βασιλεία, τότε θα μπορούσαμε να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή αυτών των χρημάτων. Γι' αυτό και από εκεί και η χρησιμότητα ορισμένων τροπολογιών και νομίζω ότι θα πρέπει να υποφεληθούμε στη συζήτηση αυτή. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε, αλλά εδώ υπάρχει μια παραπομπή σε πάρα πολλά τα οποία εξετάζονται και αφορούν τις τροπολογίες. Τρίτη σειρά τώρα παρατηρήσεων σχετικά με τους ε, οργανισμούς αξιολόγησης. Αξιολόγησης λοιπόν, γιατί θα πρέπει με τον, άλλο, με τον ένα τον άλλο τρόπο επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να φιλτράρουμε όλο το κείμενο και να δούμε αυτές τις παρατηρήσεις, πώς θα τις αφαιρέσουμε ή όχι για αυτές τις εταιρείε αξιολόγησης, αλλά θα πρέπει να έχουμε μικρότερη εξάρτηση από αυτές τις εταιρείε αξιολόγησης, οργανισμούς αξιολόγησης, γιατί εδώ τα πράγματα μπερδεύονται μετά και να εφαρμοστούν όπως πρέπει σχετικά με τη Βασίλεια. Και ακόμα δεν είπε τίποτα για το κύριο χρέος ο εισηγητής. Νομίζω ότι αποτελεί σημαντικό πάντα σημείο για το πώς ενσωματώνονται όχι αυτά στον όλο υπολογισμό και με ποιο τρόπο για μια, ένα κατάλληλο υπολογισμό για να μπορέσει να, ε, ε, να χρησιμεύσει πραγματικά αυτό το κείμενο να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Κάρας. Προφανώς το ζήτημα αυτό είναι δύσκολο και πολύπλοκο. Θα είμαι σύντομος πάντως, όπως το πες και εσύ Ότμαρ, δεν πρέπει εδώ πέρα να έχουμε ένα κατάλογο προθέσεων, προσδοκιών για τα κράτη-μέλη. Πολύ σωστό αυτό. Από την άλλη όμως λες ότι πρέπει να σταθεροποιήσουμε την εσωτερική αγορά, δηλαδή πρέπει να πετύχουμε μια ισορροπία. Πολύ συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Προτείνουμε λύσεις για τα πάντα. Θέλουμε να εναρμονίσουμε τα πάντα, παντού στην Ευρώπη. Δεν θα σταθεροποιήσει όμως κάτι τέτοιο την εσωτερική αγορά. Θα προκαλέσει αντίθετα προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη αυτά στη συνέχεια θα πειράσουν άλλα κράτη-μέλη με τη σειρά τους. Επομένως, το είπατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε, η ελαστικότητα τελικά, η ευελιξία, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον ορισμένοι ζητάμε. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο καλύπτεται σε κάποιες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι ε, αν δεν καλυπτόμαθα όμω όλοι και δεν είμαστε ικανοποιημένοι, τότε θα πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα και τι συμβαστικέ τροπολογίε και θα είμαστε έτσι πιο ικανοποιημένοι ορισμένοι. Γιατί για μένα, για τη δική μου χώρα, το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όπω η Ισλανδία. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σαν την Ισλανδία. Πρέπει επομένω να έχουμε το απαραίτητο επίπεδο προστασίας και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να προστατεύουμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Ελίσσα. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είναι τεράστιο το έργο και σας συγχαίρω για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ε, ε, τις διαπραγματεύσεις. Πολύ σύντομα για κάποια σημεία. Είναι σημαντικό το ότι λαμβάνετε υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σας ευχαριστώ που έχετε συμπεριλάβει εν μέρει και τη δική μου τροπολογία. Για τα ΣΥΦΙΣ νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Με ανησυχεί κάπως η εθνική διάσταση γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς βέβαια μας, λείπει κάποια, μας λείπουν κάποια βασικά νομοθετικά κείμενα τα οποία δεν έχουν προκύψει και αφήνω κατά μέρος το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ή κάποιου άλλου θεσμικού φορέα που θα αντισταθμίσει τον κίνδυνο για την εσωτερική αγορά και πάλι Χαιρετίζω αυτά τα οποία έχετε συμπεριλάβει, αλλά θα ήθελα μια κίνηση προς την κατεύθυνση του καλύτερου ελέγχου ε, της κυκλικότητας, του φιλοκυκλικού χαρακτήρα. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επίσης στις συνέπειες ε, των κρατικών ενισχύσεων. Οι τροπολογίες μου 1462 και 1452 προσπαθούν ακριβώς να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Όταν μιλάτε για ευελιξία και αναγνώριση επιχειρηματικών μοντέλων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πρόβλημα ε, των συμμετοχών μειοψηφία που σε μερικές χώρες ε, είναι σημαντικό ζήτημα. Και από πολιτικής πλευράς θεωρώ πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε μια ξεκάθαρη γραμμή βάσει της πορείας που έχετε χαράξει τα θέματα των αποδοχών και τα θέματα της φοροαποφυγής. Γι' αυτό το λόγο στην οδηγία θα ήθελα να ξαναδείτε την τροπολογία μου 44 για την αναφορά δεδομένων αναχώρα, γιατί αυτό νομίζω ότι θα μας προσφέρει πολλά στον τομέα της φοροαποφυγής. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας συγχαίρω για άλλη μια φορά για το έργο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλους εγγεγραμμένους στον κατάλογο ομιλητών και θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μήπως έχει να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ότμαρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο είναι μια συζήτηση υψηλής ποιότητας και αυτό αποτελεί και προϋπόθεση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα αφού όλοι έχουμε και την καλή βούληση. Είναι μια συζήτηση ε, συλλογικής ευθύνης και συλλογικής ανάληψης ευθύνης σε μια εποχή κρίσης. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεργασία και για τα σχόλιά σας. Δεν έχω ξεχάσει, επίτηδες δεν ανέφερα ε, όλα τα σημεία. Περιορίστηκα στα πέντε σημεία ε, των συμβιβαστικών τροπολογιών. Δεν έχουν κλείσει βέβαια οι συμβιβαστικές λύσεις είναι μία ενεξελίξη διαδικασία. Ακόμη επεξεργαζόμαστε αυτά τα συμβιβαστικές τροπολογίες για να ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες από τις τροπολογίες σας. Είμαστε ανοιχτοί και ανάλογα με τις περαιτέρω συζητήσεις θα υποβληθούν τελικές προτάσεις. Στόχος είναι να γίνει αποδεκτό το συνολικό πακέτο από τις πολιτικές ομάδες. Και χθες υποσχεθήκαμε ότι η γραμματεία και οι συνεργάτες μου θα καταστρώσουν ένα χρονοδιάγραμμα με όλες τις ημερομηνίες που συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις αυτές για να ξέρουμε πώς διαρθρώνονται αυτές οι προτάσεις μεταξύ τους για να υπάρχει μία συνέχεια σε όλα όσα κάνουμε. Ένα σημείο που δεν συζητήσαμε είναι αυτό το σχετικό με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις Θέλουμε να συζητήσουμε τα θέματα της πείρας που έχουμε με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις με στόχο να καταλήξουμε σε μια ενιαία θέση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία θέση που θα οδηγήσει σε προβλήματα στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να έχουμε μια ενιαία θέση που θα οδηγήσει σε μια καλή αποδοχή από το Κοινοβούλιο. Το θέμα των φυσικών προσώπων που ε, αναφέρατε εσείς το συζητήσαμε χθες. Είναι θέμα και ορισμού Έχουμε βάλει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είπαμε ότι είναι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και φυσικά πρόσωπα. Λαμβάνουμε υπόψη την ίδρυση των επιχειρήσεων και ενδεχομένως και την τροποποίηση του καθεστώτος της επιχείρησης. Και το θέμα της αγοράς ακινήτων και των στεγαστικών εταιριών επίσης μας απασχόλησε και η συζήτηση της μέγιστης και ελάχιστης εναρμόνισης. Θα θέλαμε να έχουμε στο δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση στην εσωτερική αγορά, αλλά δεν πρέπει να τα εναρμονίσουμε όλα. Χρειαζόμαστε ευελιξία. Και θέλουμε να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη έναντι των άλλων υπήρων και τις διαφορετικές τραπεζικές δομές που υπάρχουν. Αυτά σε όλα όσα αφορούν τη Βασιλεία 3. Η ευέλικτη αντιμετώπιση δεν ε, ε, μειώνει τα μέτρα τα οποία θέλουμε ε, να λάβουμε, αλλά μας δίνει διαφάνεια ε, και επιτυγχάνει ταυτόχρονα αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχει ε, κάτι το αδιαφανές πίσω από κλειστές πόρτες. Οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ευελιξία, αλλά όχι εις βάρος της εσωτερικής αγοράς. Η διαφοροποίηση λοιπόν και η ευελιξία είναι παράγοντες στους οποίους πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι σημειώνουμε πολύ καλή πρόοδο. Προφανώς πρέπει να βρεθούν και άλλες συμβαστικές λύσεις. Πάντως μέχρι στιγμής έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο. Ακολουθούμε πιστά το χρονοδιάγραμμα, το οποίο μας έχει υποδείξει ο εισηγητής. Μπορώ να κλείσω στο σημείο αυτό τη συνεδρίαση. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο στις 7 ε, το βράδυ, 17 Απριλίου. Ευχαριστώ.